Chers collègues, nous allons commencer nos travaux. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Mes chers collègues, αγαπητοί συνάδελφοι, την Παρασκευή 7 Απριλίου είχαμε μια νέα τρομοκρατική επίθεση σε μία από τις πιο όμορφες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στη Στοκχόλμη. Χρησιμοποιήθηκε ένα φορτηγό, τέσσερις νεκροί, πολύ τραυματίες. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς ε, τη φρικαλότητα, τη βαρβαρότητα αυτή. Ούτε για να εκφράσει επαρκώς ε, τη θλίψη που νιώθουμε όλοι δύο εβδομάδες αφού Εορτάσαμε εντό αγωγικών. Θυμηθήκαμε την επέτειο των ένα χρόνο της επιθέσεις ε, των ε, Βρυξελών. Ενός λεπτού σιγή παρακαλώ τη σκέψη μας σήμερα στους Σουηδούς φίλους. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ. L'ordre du jour peut être adopté. Μπορούμε να εγκρίνουμε νομίζω την ημερήσια διάταξη αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, μετακινούμε σας εκπροσωπώ όταν είμαι σε, κάποια, σε κάποιο επαγγελματικό ταξίδι. Και συγκεκριμένα για τη Μάλτα που ήμουν ε, στο Συμβουλίο θέλω να σας αναφέρω το τι συνέβη εκεί. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στη Μάλτα 28 και 29 Μαρτίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κοχ που ήταν μαζί μου. Έχουμε την κηρύξη της Βαλέτα για την οδική ασφάλεια και τις θαλάσσιες μεταφορές. Τις συζητήσαν και τις ενέκριναν στην εν λόγω συνεδρίαση. Όταν εγώ έλαβα το λόγο, περασπίστηκα ε, τα ε, συμφέροντα και της Επιτροπής μας αλλά και του κλάδου ενώπιν των Υπουργών που πρέπει να πω ότι δεσμεύτηκαν υπέρ της οδικής ασφάλειας και των θαλάσσιων υποθέσεων. Είναι σαφές ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές θέσεις ε, λήφθησαν υπόψη. Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά άμεσα το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. 26.000 νεκροί από τροχέα κάθε χρόνο. Ε, το νούμερο αυτό θα σας το επενθυμίσω. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοια νούμερα. Πρέπει οι δρόμοι μας να γίνουν πιο ασφαλείς. Να μην ισοδυναμούν με φόβο. Είμαι απόλυτα για τους ε, χρήστες. Και επειδή είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών, αλλά και πραγματική εναρμόνιση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πενθύμησα στη Μάλτα λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας Επιτροπή ιδιαιτέρως ήδη έχουν εγκρίνει ε, ψηφίσματα για την οδική ασφάλεια και στο θαλάσσιο τομέα επίσης, για τον θαλάσσιο τομέα και θα ήθελα να σας προτείνω να επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια σε κάποια μελλοντική συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών. Θα ήθελα επίσης να προσκαλέσω τον κύριο Ζάντο, που είναι ο ειδικό απεσταλμένο των Εθνών για την Οδική Ασφάλεια, να έρθει να μα ε, αναφέρει τον πολύ εντυπωσιακό, τα, τα, σχετικά με τον πολύ εντυπωσιακό λόγο που ε, εκφώνησε στη Μάλτα και θα ήθελα επίση η Επιτροπή Μεταφορών να δεσμευτεί πραγματικά, ιδίω όταν θα συζητηθεί το πακέτο των οδικών μέτρων για να αναφέρουμε τα περί της οδικής ασφάλειας αυτά. Δεν θέλουμε να έχουμε μόνο διακήρυξεις υπουργών που τις υπογράφουν απλά οι εκπρόσωποι των κρατών μελών. Πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να έχουμε πραγματικά και τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να προωθήσουμε την οδική ασφάλεια. Αυτά είχα να πω και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην κοινή συζήτηση ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, ευρωπαϊκά πρότυπα και εφαρμογή του κανονισμού 1025 του 2012. Ήτρε και ΙΜΚΟ είναι οι καθηγητές επιτροπές, εμείς γνωμοδοτούμε. Η συγητής, ο κύριος Τέλιτσκα. Καλώς ήρθατε. Να δώσω βέβαια το λόγο στον κ. Τέλης, και στους κοιόδης ηγητές, εφόσον θέλουν να λάβουν το λόγο, για τα θέματα αυτά. Και στη συζήτηση, στο τέλος της συζήτησης φυσικά θα καλέσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετηθούν, ώστε πραγματικά να ακούσουμε ε, την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ε, έχω αναλάβει δύο γνωμοδοτήσεις. Θα τι συζητήσουμε από κοινού εφόσον πρόκειται για κοινή συζήτηση. Αντικατοπτρίζει το έργο αυτό που έχω κάνει και το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν θα επαναλάβω κυρία Πρόεδρε ότι έχω προείπει στη συζήτηση που είχαμε το Φεβρουάριο. Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πώς έχει προχωρήσει η επεξεργασία των συμβαστικών τροπολογιών από εκείνο με τους γιώδες εισηγητές και ε, συνεχεία θα αναφέρω κάποιες αλλαγές. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι και το εννοώ αυτό που θα πω, ε, ότι όλοι οι εισηγητές συμμετείχαν πολύ επικοδομητικά και το βλέπουμε αυτό, ότι είχαμε 200 τροπολογίες και μέσα σε μια ώρα συνεδρίασης ε, τα καλύψαμε όλα αυτά τα θέματα και για τις δύο γνωμοδοτήσεις. Ε, ασυνήθιση ίσω η διαδικασία, αλλά επαγγελματική, επικοδομητική, όπω είπα. Και ευχαριστώ ειλικρινά του κοιόδη. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να δυσαρεστηθούν ε, βλέποντα ότι δεν έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο ευκαιριών αυτό το κάνουμε σκοπίμως, διότι νομίζω ότι έχουν κατατεθεί στο παρελθόν πάρα πολλές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε ξανά όλες τις ευκαιρίες που είχαμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω κάποια σύγκριση. Γιατί αν έκανα θα ήταν σαν να συζητώ με τον προηγούμενο αιώνα τι ε, ευκαιρίες πρόσφερε η ανακάλυψη του αυτοκινήτου, για παράδειγμα και πώς μπορέσαμε να το αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν εστιάζουμε σε κάποια επικαιρά στοιχεία και σημεία. Θέλουμε να δούμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους και δεν επαναλαμβάνουμε ένα μακρύ κατάλογο Ευχαριστώ και δυνατόν που βέβαια σίγουρα θα προκύψουν. Τρία σημεία θέλω να υπογραμμίσω. Αυτά αναφέρονται άλλωστε και στις γνωμοδοτήσεις. Και νομίζω ότι επέφεραν και μια αλλαγή σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Το πρώτο. Συμπεριλαμβάνουμε τις νοφεί επιχειρήσει και τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια αυτό ήταν στο σχέδιο γνωμοδότηση και πριν, όμως τώρα νομίζω ότι δίνουμε τη δέουσα προσοχή με τη συμβαστική πρόταση στις δύο αυτές ε, κατηγορίες επιχειρήσεων. Δεύτερον, μέσο τουρισμού. Ξετάσαμε το θέμα όχι από πλευρά των τουριστικών υπηρεσιών, αλλά είδαμε την ευρύτερη εικόνα. Το πώ δηλαδή συνδέεται ο τουρισμό με τις μεταφορές. Ψηφιοποίηση, τυποποίηση θα προσφέρουν σίγουρα πολλέ δυνατότητες. Προσπαθήσαμε να δείξουμε την αντικειμενικότητα του τομέα. Τρίτη αλλαγή, δημιουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική διάσταση. Αλλά σε σύγκριση με κάποιες ε, από τις κάποιες τροπολογίες και κάποιες απόψεις που μπορεί να είχαν κάποιοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η διατύπωση είναι θετική. Διερωτώμεθα, δηλαδή. Για την ψηφιοποίηση που μπορεί, και δεν το αρνούμε, να επηρεάσει τη θέση ε, την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να την ε, ε, σταματήσουμε για αυτό το λόγο. Δεν νομίζω. Το θέμα είναι που θα εστιάσουμε. Θα πρέπει να εστιάσουμε στους ανθρώπους και να δούμε αυτοί οι άνθρωποι που θα χάσουν τη δουλειά τους, πώς μπορούν να αποζημιωθούν. Τι εργαλεία μπορούμε να βρούμε. Αυτό είναι το αυτός είναι ο στόχος μας. Επίσης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εγκύψουμε πολύ στα θέματα της χρηματοδότηση. Τα έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν και κάποιες δυνατότητε στο μέλλον με τις υποδομέ που δημιουργηθούν. Δεν εστιάσαμε λεπτομεριακά σε αυτό το σημείο. Απλά είπαμε ότι Ξέρουμε τι έχουμε και ελπίζουμε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι κατά το του δυνατό βαθμό. Ένα άλλο θεμητό ζήτημα που δεν αναφέρεται βέβαια στη της είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όσο περισσότερο ψηφιοποιούνται οι μεταφορέ, ε, όσο περισσότερο αυτοματοποιούνται οι μεταφορέ, τόσο μεγαλύτεροι κίνδυνοι ελοχεύουν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι η σωστή θέση και η σωστή στιγμή να προβούμε σε ένα εγχείρημα ανάλυση αυτών των κινδύνων. Είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποια στιγμή θα καταρτήσει μια σύσταση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επομένως, ε, εκεί θα είναι και η κατάλληλη στιγμή να αναφέρουμε και εμείς τις δικές μας ε, απόψεις και συστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Αυτά νομίζω είναι τα όσα έπρεπε να αναφερθούν στην νομοδότηση ε, σε συνέχεια της συζήτηση που είχαμε το Φεβρουάριο και της ανάλυσης των συμβαστικών τρόπων. Σας ευχαριστώ γιατί είχαμε μια μοναδική συνεργασία και παραλαμβάνω τις φορές του Σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Τέλιτσκα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γέρκινα. Thank Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή μας, τον κύριο Τέρισκα και όλους τους και όλους εισηγητές. Ε, νομίζω ότι η ατμόσφαιρα που επικράτησε στη συνεδριάση μας ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Το είπε και ο εισηγητής και τελικά κατάληξαμε σε μια γνωμοδότηση συνεκτική και ισόρροπη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή, γιατί από πλευράς ΕΛΚ βλέπουμε ότι η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στη βιομηχανία είναι κρίσιμη για να δοθεί μια όθηση ε, στην οικονομία και στις μεταφορές φυσικά για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Και ισχύει και για τον τουρισμό αυτό. Η ψηφιοποίηση πολλές φορές προσφέρει νέες ευκαιρίες ε, για τις μεταφορές οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες ε, λειτουργούν με τρόπο πιο βιώσιμο, πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό και συχνά φθηνότερο. Είναι καλό λοιπόν που έχουμε αυτό το θετικό πνεύμα και τη θετική στάση απέναντι στην ψηφιοποίηση. Ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι ανισχύει πολύ ο κόσμος, μήπως χάσει τη δουλειά του λόγω της ψηφιοποίησης, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αλλάζει η αγορά εργασίας, αλλά ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και το ανθρώπινο δυναμικό, το εργατικό δυναμικό να προετοιμάζεται, να ε, προσαρμόζεται σε αυτό το νέο κόσμο. Και στην Ευρώπη εμείς θα πρέπει να είμαστε ηγέτες στην προσπάθεια αυτή και στη διαδικασία. Είναι πολύ ισορροπημένη λοιπόν και θετική η γνωμοδότησή μας. Δύο λόγια για τα πρότυπα. Αν κατάλαβα καλά, αναφέρθηκε και στην άλλη γνωμοδότηση ο κύριος Τέλητσκα, για τα κοινά πρότυπα είναι μια σημαντική βάση έτσι ώστε να δρέψουμε όλους τους καρπούς της ψηφιοποίησης στην ενιαία αγορά και είναι σημαντικό η Ευρώπη να ε, επιζητεί ε, πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιούνται διεθνώς. Να έχουμε νέες υπηρεσίες κινητικότητας, νέες καινοτομίες στις μεταφορές και ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη δική μας γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών θεωρούμε ότι είναι πραγματικά πολύ ισόρροπη και αυτή η ε, γνωμοδότηση. Ευχαριστώ τον Παύελ Τέλιτσκα και όλους τους υπολείπους και όσοι ιδέες. Νομίζω ότι εργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά και γόνιμα και οι αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές να τις βρουν χρήσιμες. Καμιά φορά είναι δύσκολα τα χρονοδιάγραμματα, γιατί επί της ουσίας αρμόδιες επιτροπές ε, συντάσσουν τις, επιτρο... Ε, ε, τροπολογίες του συγγνώμη, ταυτόχρονα με εμά. Οπότε για να πιάσει τόπο η γνωμοδότηση μιας επιτροπής όπως η Επιτροπή Μεταφορών ίσως χρειάζεται να ξαναδούμε τα χρονοδιαγράμματα. Βέβαια αυτό μπορεί έχει να κάνει και με τις διακοπές του Πάσχα, πάντα πιέζει ο χρόνος σε τέτοιες περιστάσεις. Ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία. Euh, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Ουγγελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Τέλιτσκα, ολοκληρώσαμε μια δουλειά συναρπαστική και πολύ ενδιαφέρουσα και τα αποτελέσματα νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά. Όταν μιλάμε για το μέλλον, οι, οι εμπειρογνώμονες και ευρωβουλευτέ ειδικοί στου διάφορου κλάδου που συζητήσαμε μπορούν να έχουν διαφορετικέ απόψει για τι διάφορε προκλήσει που έχουμε μπροστά μα. Συμφωνώ και το ανέφερε και ο κ. Στέλιτ αρκετέ φορέ. Είμαστε ε, ε, στα μέσα μια πλήρου διαδικασία νέα βιομηχανοποίηση μια βιομηχανική επανάσταση. Αν δούμε τι είχε γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχε καταστάσει, βλέπουμε ότι δεν ε, άγγιζαν οι επαναστάσει αυτέ ένα μόνο βιομηχανικό κλάδο, αλλά επηρέαζαν κάθε είδου δουλειά και επηρέαζαν δομικά την διοργάνωσή τους. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερα υπεύθυνη στάση ε, ως προ τις αλλαγές αυτές στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω η γνωμοδότηση του κυρίου Τέλιτσκα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τέτοιου σεβασμού προς την... και επίγνωση προ τι αλλαγέ που συντελούνται. Εγώ ξέρω περισσότερα για τον κλάδο του τουρισμού και ευχαριστώ τον κύριο Τέλιτσκα που δέχτηκε τι προτάσει μου. Αναφέραμε και τι ε, βιομηχανίε δημιουργικέ που είναι σημαντικέ για όλου μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πολύ ποιοτική γνωμοδότηση για τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Να πω ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ απλό, εύληπτο σύστημα προτύπων που να μπορεί να χρησιμοποιείται απλά και να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών αγορών, χωρίς περιττό διοικητικό άχθους, με ευκολία. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για να είμαστε πλήρως από... προετοιμασμένοι για τη νέα βιομηχανική επανάσταση. Στηρίζουμε τις προτάσεις σας και θέλω να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους και όλους εισηγητές, αλλά όλος ιδιαίτερα τον κύριο Τέλιτσκα για την πολύ καλή δουλειά που έγινε. Με μεγάλη χαρά να ξανασυνεργαστούμε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Ζήλε δεν είναι εδώ. Το λόγο έχει λοιπόν η κυρία Κιλόνεν. Παρακαλώ κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον γιατί τον κύριο Τέλητσκα. γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας. Ω και ό,τι συγκέντρια πρέπει να πω ότι ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η τυποποίηση και η ταχεία ψηφιοποίηση το διαδίκτυο των πραγμάτων που χρειαζόμαστε τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, όλα αυτά τονίζονται με τον σωστό τρόπο στην έκθεση αυτή. Πρέπει να συνεχιστούν οι αλλαγές και εμείς να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, να έχουμε επίσης έναν ευπροσάρμοστο τουριστικό κλάδο στην Ευρώπη. Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκθεσης είναι ότι οι πληροφορίες έχουν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία στο σχεδιασμό των συστημάτων και δικτύων μεταφοράς έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες όσο το δυνατόν περισσότερο με ευφυείς ε, εφαρμογέ για τα κινητά και τέτοιου είδους τεχνολογικές λύσεις που να μας δίνουν περισσότερες δυνατότητες. Από την άλλη βέβαια πρέπει να προσέξουμε οι διεπαθές και τα αρχεία δεδομένων που τηρούνται να είναι ασφαλή. Πρέπει να δώσουμε και τα ανάλογα κίνητρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να προσφέρουμε ευκαιρίες ψηφιοποίησης και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα ισχύσει για τις μικρομεσαίες, γιατί είναι σημαντικό να έχουν βελτιωμένη πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Πολλά από τα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δαπανηρά ε, και ακριβά οι διαδικασίε πρόσβαση είναι ακριβέ αν το δει κανεί από το πρίσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά από εμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κιλόνεν. Από τους πράσινου ο κύριος Τέιλορ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον είστε παρατηρητικοί, θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν είμαι η έχει καθυστερήσει, αλλά μου έστειλε το σημείο της για να το διαβάσω. Και για τις δύο αυτές εκθέσεις. Η ψηφιοποιημένη ευρωπαϊκή βιομηχανία και η σχετική έκθεση παρουσιάζει πολλές προκλήσεις όπως και ευκαιρίες, ιδίως στον τομέα των μεταφορών. Η κυρία Evans θεωρεί ότι η έκθεση του κυρίου Τελίτσια καλύπτει κάποιες από αυτές τις ε, προκλήσεις και κάποια τα προβλήματα για τις ενδεχόμενες αλλαγές στην κοινωνία έχει συντάξει τροπολογίες ε, για την ε, ψηφιοποίηση και την αποτίμησή της επίσης ε, και για τη βιωσιμότητα και χαίρεται που θα απηχηθούν στην έκθεση. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη σχετική έκθεση, η κυρία Εβανς θεωρεί ότι το κείμενο των συμβαστικών λύσεων είναι πολύ ισόρροπο και χαίρεται ιδιαίτερος που συμπεριλαμβάνονται κάποιες από τις δικές της τροπολογίες Ιδίω οι αναφορέ στι κλιματικέ αλλαγέ, τον τουρισμό, την διαλογικότητα και την ευκολία τη πρόσβαση. Ευχαριστεί λοιπόν θερμά τον εισηγητή και με μεγάλη χαρά θα στηρίξει πλήρω και τι δύο εκθέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τέ. Μην ανησυχείτε, δεν σας μπέρδεψα με την κυρία μας. Σας το υπόσχομαι, δεν πρόκειται να το κάνω. Συνεχίζουμε κυρία Γιώτο. Με συγχωρείτε κυρία Ντανάτο. Α, δεν είναι εδώ. Η Αυτιντή έχει κάποιον άλλο που θα πάρει το λόγο. Δεν είναι εδώ η συνάδελφός μου, αλλά δεν μου έδωσε και τις ε, σημειώσεις της για να τις διαβάσω. Τέλεια. Συνεχίζουμε με τους συναδέλφους. Ο κύριος Βάντεν Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Βίρκουνεν, συνάδελφός μου του Λαϊκού Κόμματος. Έχω ενοχληθεί κάπως από το γεγονός ότι εμείς κάνουμε εδώ γνωμοδοτήσεις και οι αρμόδιες επί επιτροπές έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο τους και από δημοκρατική σκοπιά να το δείτε είναι άκρος ε, προβληματικό αυτό. Θα το θέσω και στη συνεδρίαση των συντονιστών όπου θα επανέλθω. Θα πρέπει κάπως να συντονίζουμε ε, και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας με τις άλλες επιτροπές γιατί αλλιώς αυτό είναι φλιβερό ε, και καταθλιπτικό. Δηλαδή κάνουμε εμείς νομοδότηση και πάει στο βρόντο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή, κύριε Βάντεν Κάμπ. Κύριε Ντερμόντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον σκιώδη εισηγητή, του εισηγητή μάλλον και τους σκιώδη εισηγητέ για τη δουλειά του, και του ευχαριστώ που συμπερίλαβαν το τμήμα που αφορά τον τουρισμό κάτι που θα ήταν ε, αμέλεια εκ μέρου μα να μην το συμπεριλάβουμε όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα θέματα. Ε, επί τη ουσία η Επιτροπή μα έχει και αυτή την αρμοδιότητα, οπότε πρέπει να εργάζεται για να επιτυχάνει τα σωστά αποτελέσματα. Ήθελα λοιπόν να δοθεί έμφαση σε ορισμένα από τα περιεχόμενα της έκθεσης, δεν μπορεί να διευκριστεί ότι ω προς τον τουρισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατηρεί την όθηση τη ε, δημιουργική βιομηχανία, όμω η γνωμοδότηση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να καλύψουμε και αυτόν τον κλάδο. Και χρειάζεται και μια ε, νομοθετική διευθέτηση που να είναι προσαρμοσμένη στι νέε τεχνολογικέ λύσει. Δεν μπορούμε να προβλέπουμε νομοθετήματα που να είναι εκτό τη σημερινή πραγματικότητα, αλλά να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Και επίση, παρά το γεγονό ότι πρόκειται αρμοδιότητα, για αρμοδιότητα τη ΣΥΜΚΟ, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη προστασία των καταναλωτών ακόμη και σε ό,τι αφορά τους τίτλους ταξιδιών, διότι όλο και περισσότερο θα υπάρχουν πλατφόρμες που θα προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ταυτόχρονα όμως και εμείς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι καταναλωτές προστατεύονται σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και διαλογικότητας των διαφόρων συστημάτων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ανεμπόδιστα τα δίκτυα μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρέφομαι μέσα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όρες γνωμοδοτήσεις. Και είπαν και όλοι οι σκιώδεις ηγητές ότι ο κύριος Τέριτσκα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουμε όλοι κοινό στόχο. Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και επανάστασης μάλιστα της ψηφιακής εποχής, θα πρέπει να δούμε πώς επιδρά αυτό στις επιχειρήσεις μεταφορών, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτίθεται να πράξει, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με βάση ποια νομοθεσία. Ε, ακούσαμε για ψηφιακές πλατφόρμες, που είναι ένα θέμα το οποίο συζητούν τα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο. Στον κύριο Κονζάλε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είστε εδώ, πού είστε, σηκώστε το χέρι σας. Γεια σας, καλημέρα. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Εμίλιο Κονζάλε από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις που είναι. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές στο συντακτηνομοδότηση που εξέτασαν το θέμα αυτό από τη σκοπιά των μεταφορών ε, και την ψηφιοποίηση και την τυποποίηση. Καμιά φορά ακούμε επικρίσει στην γνωμοδότηση για το γεγονός ότι έχουμε επικεντρωθεί στην ε, ε, δική μας γενική διεύθυνση για το πώς θα ρυθμίσουμε την ηλεκτρονική κλίση, το περίφημο e-call. Αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει μόνο, αλλά γενικότερα ψηφιοποίηση, ψηφιακή καινοτομία και άλλοι τομεί των μεταφορών. Η ψηφιοποίηση, ε, η πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση στην ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία αφορά ε, όλη τη διαδικασία της παραγωγής, εφοδιαστικής μεταφορών, προϊόντων και υπηρεσιών. Όλοι αυτοί θα υποφεληθούν και υπάρχει δυνατότητα ε, νέων επιχειρηματικών μοντέλων ε, και νοτόμων που ζητούν και οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες έτσι ώστε ο κλάδος αυτός να τοποθετηθεί καλύτερα και σε πιο ανταγωνιστική θέση στη διεθνή κονίστρα προωθώντας ε, και τις θέσεις ε, εργασίας και την ανταγωνιστικότητα. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν από τη Γενική μας Διεύθυνση. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή, έχουμε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας και πιστεύουμε ότι ο κλάδος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να υποφεληθούν και να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο παγκοσμίως. Σε αυτό συμφωνούν πολλοί ενεχομένοι, τους οποίους ρωτήσαμε πρόσφατα. 27 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει και άλλα δύο ε, μέλη ΕΖΕΣ για να υποστηρίξουν ε, διαδρόμους για τα αυτόματα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Επαναλαμβάνω όμω δεν είναι αυτό ε, που μας απασχολεί και δεν έχει συγκεντρώσει όλη μας την προσοχή το θέμα των οδήγηση της οδήγησης αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Ε, έχουμε και άλλες ε, κατευθύνσεις όπως αυτές που αναφέρει ο εισηγητής νέες εταιρείε, νεοφυείς, μπορεί να κλείνουν κάποιες μικρομεσαίες, ανοίγουν κάποιες άλλες, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Και όπως σας είπα προηγουμένως, και ο τουρισμός είναι σημαντικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση εκεί. Και όπως σας είπα, η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι διακλαδική. Δεν αφορά ένα και μοναδικό κλάδο και φυσικά και τις μεταφορές και τον τουρισμό. Και τέλος, για τα πρότυπα, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι ό,τι έχει ε, να κάνει με διασυνδεμένα αυτόματης οδήγηση αυτοκίνητα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρακολουθήσει εξελίξεις, ε, την έρευνα, τα αποτελέσματα και τα διεθνή πρότυπα και ε, η διασφάλεια στον κυβερνό χώρο που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο τα διασυνδεδεμένα και αυτόματης οδήγηση αυτοκίνητα. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κονσάλες, ακούσαμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Βαντενκάμπ, προς ενημέρωσή σας, ακόμα και να έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε στους συντονιστές, για τις ψηφοφορίες. Στην Ήτρε θα ψηφίσουν στις 24 Απριλίου σε 15 μέρες και στην Ήμκο ανέβαλαν την ψηφοφορία. θα ψηφίσουν το Μάιο. Πράγμα που αφήνει κάποιο χώρο στην Επιτροπή μας και κυρίως στον εισηγητή για να επηρεάσει την έκθεση και της Επιτροπής Βιομηχανίας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Εσείς πάντως έχετε, κύριε Τέλιτσκα, όλη την υποστήριξή μας και τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, εκτιμώ αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Μας επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με καθυσυχάζει λίγο γιατί είχα ανησυχήσει ότι τα διασυνδεδεμένα οχήματα και τα αυτόματα οδήγηση χωρί οδηγό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα πολύ πιο σημαντικά και επίγοντα. Και για τον τουρισμό ε, και τις μεταφορές δεν είναι μόνο δύο χωριστά πράγματα, αλλά υπάρχει αλληλοδιείσδυση. Ε, υπάρχουν ε, μεγάλες διασυνδέσεις μεταξύ τουρισμού και ε, μεταφορών και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν έχουμε συμβιβαστική τροπολογία για να το διευκρινίσω αυτό. Ήταν η δική μου τροπολογία υπαριθμών 57 ε, που γνώρισε μεγάλη υποστήριξη συνενετικά από όλους τους συναδέλφους για τις δύο γνωμοδοτήσεις. Μία τροπολογία πρέπει να ψηφίσουμε χωριστά. Δεν θα ακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέλη. Τσικά ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο το πρωί, 9 το πρωί συγκεκριμένα. Ελπίζω να το σημειώσατε στις ατζέντες σας και τώρα συνεχίζουμε περνώντας στο επόμενο σημείο την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς οι απόλυμες των ατόμων της κοινότητας κτλ. Κυρία Μπιλμπάο είναι η συγγήτρια. Θα λάβω πρώτο λόγο και εν συνεχεία οι σκιώδεις εισηγητές και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα έχει μέχρι τότε ακούσει. Κύριε Μπιλμπάου, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήδη στο Στρασβούργο ε, είχαμε μία συνάντηση με τους χιώδες εισηγητές. Πέντε συμβαστικές προτάσεις ε, κατατέθηκαν, ε, των οποίων οι τέσσερις αφορούν την προστασία δεδομένων. Υπήρχε και μία ανησυχία από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και επίση και από την κυρία Μοντέρο Αγγιλιάρη είχαμε ακούσει μια αντίστοιχη ανησυχία. Δηλαδή όταν ε, θα πρέπει αυτές οι πληροφορίε να διαγράφονται αυτόματα ή άμεσα, αμελητή. Έπρεπε να δούμε ποια από τις δύο λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε. Είχαμε διαβουλεύσεις ε, και με τους γλωσσομαθείς νομικούς Καταλήξαμε σε μία πρόταση λοιπόν, όπου λέμε τελικά ότι θα πρέπει να ε, διαγράφονται αυτόματα οι πληροφορίες χωρίς αχρίαστη καθυστέρηση, λέμε. Και πιστεύω ότι έτσι καλύπτονται οι ανησυχίες και της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ευθεριών ΛΥΜΠΕ αλλά και της ε, Βουλευτού του ΕΛΚΑ. Πέμπτη, ε, συμβαστική τροπολογία έχει να κάνει με την ενσωμάτωση, τη συμπερίληψη της πληροφορίας για την ηθαγένεια του ατόμου. Αλλά αυτή η ε, συμπερίληψη της πληροφορίας θα είναι εθελοντική, ε, οθελή. Νομίζουμε ότι δίνει πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν για τη διάσωση, για την οικογένεια που θα ενημερώνεται και για τις δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν αμέσως μετά από κάποιο ατύχημα. Εν γέννη τώρα να πω ότι από ό,τι μας είπαν στις πολιτικές ομάδες και οι σκιώδεις υπάρχει συνένεση σε μεγάλο βαθμό. Φυσικά θα ακούσω πολύ προσεκτικά και σήμερα τι θα πούν οι συναδελφοί μου για να δω αν υπάρχει ακόμη αυτή η συνένεση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπιλμπάου. Η κυρία Μοντέρο είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για τη συνεργασία τους σε αυτό το ντοσχέ. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία όλοι και όπως είπε η συνάδελφος Μπιλμπάου, ε, υποβλήθηκαν 78, συμβαστικές, 78 ε, τροπολογίες με 5 συμβαστικές λύσεις και ήθελα εδώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα στηρίζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα που θα πρέπει να εγκρίνεται από το κάθε κάτω μέλος, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τους μικρούς φορείς. Επίσης, παρόλο που πιστεύουμε ότι το μέλλον περνά από την έγκριση της υλοποίησης της ενιαίας Ευρωπαϊκής Στηρίδας, σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτή η πραγματικότητα δεν είναι ακόμη αρκετά προχωρημένη. Δεν έχει υλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά το ένατο άρθρο που αναφέρεται στην τροπολογία 78 και αφορά τα ταξίδια μικρής διάρκειας με την εξαίρεση αποστολής πληροφοριών για ε, διαδρομές διάρκειας μικρότερης της μιας ώρας. Εκεί η αποστολή πληροφοριών συνεχίζει να είναι υποχρεωτική αλλά επιτρέπεται μια περισσότερη ευελιξία ζωτικής σημασίας για κάποιες ε, θαλάσσιες διασυνδέσεις μεταξύ νήσων ως προς τα 10 λεπτά για την αποστολή των πληροφοριών και την ε, προθεσμία αυτή έγινε μεγάλη συζήτηση και βεβαίως εδικαιωδεται η ασφάλεια των επιβατών, όμως στην πράξη έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Αμφιβολίες σχετικά με τους υπεύθυνους φορείς. Θα είναι σε θέση να δώσουν αυτή την απάντηση εγκαίρως και ορθώς όπως προτείνεται. Διότι παρόλο που μιλάμε για σύστημα ψηφιοποίηση και θέλουμε να υπάρξει αυτοματοποίηση, εδώ πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε μην ε, χρησιμοποιούμε διπλά τους ίδιους πόρους και χρησιμοποιούμε αυτή τη, αυτό το διάβλο για να στέλνουμε δύο φορέ τι ίδιε πληροφορίε. Επίση, για του δύο μήνε προβλέπονται κατά κάτι μέλη για την υλοποίηση αυτή τη πρόταση είναι πολύ μικρή η προθεσμία. Γι' αυτό εγώ πρότεινα του 24 μήνε όπως αναφέρεται και στην τροπολογία 85. Όμως, κατά τα άλλα, να πω ότι ήταν πραγματικά επικοδομητική η συζήτηση και ο διαλογός μας και μπορέσαμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές λύσεις με μια έκθεση που πιστεύω ότι είναι θετική. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μοντέρο. Ο κύριος Σούλου είχε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητά για την γνωμοδότηση. Έχουμε συνεργαστεί εξαιρετικά μεταξύ μας και καταφέραμε να συνεδριάσουμε αρκετές φορές ε, και συζητήσαμε εκεί όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι ε, καταφέραμε να απαλείψουμε οποιαδήποτε άλλη επικάλυψη. Η καταγραφή λοιπόν ε, τώρα των επιβατών γίνεται με πολύ αποκλεισματικό τρόπο και αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί τώρα είναι ποιο χρειάζεται την ενιαία θηρίδα και ποιο χρειάζεται το αυτόματο σύστημα αναγνώριση για την ε, ε, διαβίβαση δεδομένων. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικέ λεπτομέρειε. Τα συζητήσαμε πάντω αυτά τα θέματα και εμεί, από πλευρά Σοσιαλιστών Δημοκρατών στηρίζουμε και τι ε, ε, τρεις συμβαστικέ προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές γιατί είμαστε πολύ ε, ικανοποιημένοι από την γρήγορη ε, και αποτελεσματική μας συνεργασία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις προτινόμενες αλλαγές που αφορούν την προστασία δεδομένων, την υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών και τις ε, διάφορες ε, ε, τροποποιήσεις ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά στις νησιωτικές περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Μπιλμπάου Ήμουν την πρώτη εβδομάδα στο Στρασβούργο Συνδριωστών των Ασκιωδών Συγητών και χαίρομαι εκ μέρου των Πρασίνων που μπορώ να σας αναφέρω ότι στηρίζουμε όλες τις βασικέ προτάσεις τις οποίες συμφωνήσαμε στο Στρασβούργο. Το βασικό για εμά, αυτή την έκθεση ήταν να εξασφαλιστεί η προστασία δεδομένων για τους επιβάτες των πλοίων και των σκαφών. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία ώστε τα δεδομένα των επιβατών να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ε, ασφάλειά του. Και βέβαια εφόσον τηρείται και η ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης. Χαιρόμαστε λοιπόν που βλέπουμε να έχετε συμπεριλάβει το θέμα αυτό και περιμένουμε με υπομονησία την ψηφοφορία όπου και θα στηρίξουμε την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Τέιλορ. Τώρα να δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλημερίσω την κυρία Κόσεμψκα από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΟΥΒ που έχει ξανάρθει στην Επιτροπή μας. Έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να καλώ, καλησπέρισω και εγώ όλους τους συμμετέχοντες. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρα και τους χειώδεις εισηγητές για την πολύ εντατική δουλειά που έκαναν ε, πάνω στην έκθεση αυτή. Καλωσορίζουμε το έργο που έχει τελειώσει μέχρι στιγμής κάποια σχόλια σε σχέση με ό,τι ε, μόλις υπόθηκε και τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουν ως στόχο τη διευκρίνηση ε, του τι θα γίνεται με τα δεδομένα τα οποία ε, διαβιβάζονται. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που γίνεται αυτή η διευκρίνηση με το χωρίς αχρίαστη καθυστέρηση. Είναι καλή έκφραση αυτή. Επίσης, ε, για πιο σύγχρονου τρόπους επικοινωνίας, ηλεκτρονικά συστήματα, υπάρχουν και τροπολογίε, υπάρχει η διακήρυξη τη Λαβαλέτα, ήταν και πρόεδρο εκεί στη Μάλτα πριν από δύο εβδομάδε, οπότε και συζητήθηκε το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη φαίνεται να θεωρούν σαφή την ανάγκη ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών συστημάτων για τη διευκόλυνση ανταλλαγή πληροφοριών στο θαλάσσιο τομέα. Σημειώνουμε επίση τι τροπολογίε, οι οποίες εξετάζουν πιο πολύ το θέμα της ε, πιο σύντομης προθεσμή για την υποβολή δεδομένων ε, των επιβατών. Πρέπει να γίνεται γρήγορα αυτή η ανταλλαγή, η διαβίβαση δεδομένων, πρέπει να υπάρχει ισορροπία, να υπάρχει ένας χρόνος επαρκής ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι σωστά αυτά τα δεδομένα. Και ένα ακόμη σχόλιο γιατί και Κίλον και ο κύριος Τέιλορ, μίλησαν για τα προσωπικά δεδομένα. Πράγματι, οτιδήποτε γίνει σε σχέση με την διεύθυνση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ε, της οδηγίας θα γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση προς ε, τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ούτως ή άλλως θα ίσχυαν οι σχετικές διατάξεις. Το λέει η Επιτροπολή, για τέλος πάντων το Αναγνωρίζουμε, ε, ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα για το Κοινοβούλιο πάντοτε και λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη τη σχετική τροπολογία και τα σχόλια των ε, εισηγητών. Για την επόμενη δεν το παραλαμβάνω, το λέω ε, για αυτήν, ότι φυσικά και θα συνεργαστούμε με όλους εσάς στα επόμενα στάδια και σε συνεργασία με το Συμβούλιο για την ολοκλήρωση των τριών προτάσεων που αφορούν ε, την ασφάλεια των ε, ε, επιβατηγών πλοίων. Είναι μια προτεραιότητα της Μαλτέσκης Προεδρίας. Βλέποντας την προσέγγιση που ακολουθείτε, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την θετική έκβαση αυτών των τριών προτάσεων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την εκπρόσωπο της Επιτροπής και τώρα να δώσω και ξανά το λόγο στην συγκήτρια μας, στην κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ όλες τις ε, πολιτικές ομάδες για τη θετική και επικοδομητική συνεργασία τους. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους υπαλλήλους που μας βοήθησαν έτσι ώστε να εγκριθεί η έκθεση με τέτοια ευκολία και να είναι και τέτοια ποιότητας. Εγώ δεν μπήκα σε λεπτομέρειες τροπολογιών, τα έχουμε συζητήσει αυτά στη συνεδρίαση των σκιωδών. Περιορίστηκα στις ε, συμβαστικές τροπολογίες και τα πιο επίμαχα. Τώρα όμως θέλω να απαντήσω και σε κάποιες ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις τροπολογίες 17 και 18 θα τις αποσύρουμε. Έχουμε εξηγήσει γιατί. Δεν θέλουμε να μειώσουμε τις προθεσμίες σε σχέση με όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλύσει τις εξαιρέσεις μας είπαν ότι δεν τους αρκεί ένα τρίμηνο, αλλά το αποφασιστικό στοιχείο ήταν το εξής. Αν δεν μπορούσαν να λύσουν διαδικαστικά αυτό το θέμα εντός τριμήνου, θα υπήρχαν προβλήματα με το ψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι λεπτομέρειε. Δεν τα ανέφερα προηγουμένω. Τα έχουμε συζητήσει με του κοιόδη. Απαντώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τις συμβαστικές. Μιλούμε επίσης και για τους χρόνους διαβίβασης των πληροφοριών. Τα 30 λεπτά όταν πρόκειται για τέτοιες πληροφορίες που ε, αυτόματα και άμεσα συλλέγεται, είναι υπερβολικό. Γιατί έχουμε διαδρομές ε, με επιβατικά πλοία που διαρκούν μία ώρα. Δηλαδή χρειάζεται μισή διαδρομή για να διαβάσει στοιχεία επιβατών. Ξέρουμε πως τα 10 λεπτά ήταν πιο σκόπιμο και πιο λογικό διάστημα. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες το βρήκαν λίγο. Αλλά για μας 30 λεπτά είναι πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ε, και απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις πολιτικές ομάδες και στην κοινή λογική. Ε, θα είναι καλή έκθεση, είμαι βέβαια, γιατί όλοι κατέβαλαν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπελμπάου. Θυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί από τις 9 και μετά. Ε, συνεχίζουμε. Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ρορό και ταχύπλο επιβατηγά σκάφη. Η συγκητή μα είναι ο κύριο Ρικέ, στον οποίο και δίνω μέσω στο λόγο και μετά οι σκιώδεις συγητές και θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στις ερωτήσει. Παρακαλώ, κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους σκιώδες εισηγητές. Στα πλαίσια του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη ρύθμιση και το θετήν, το Better Regulation, για μια έκθεση που τροποποιεί μια οδηγία και καταργεί μια άλλη. Είναι αρκετά τεχνική η έκθεση αυτή. Πώς τη δικαιολογεί. Γιατί χρειάζεται ειδική ρύθμιση τα συστήματα επιθεωρήσεων με τα ferry Όλοι σας έχετε πάρει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας, αν όχι περισσότερο, ένα ferry bot. Και ξέρετε πώς φορτώνονται τα αυτοκίνητα. Ε, κυρίως ε, ε, γίνεται από την πλώρη ε, και όταν υπάρχουν προβλήματα, ε, ναυάγια και δράματα είναι πάρα πολύ εκτεθειμένα. Θυμάστε τι είχε γίνει στη Σουηδία, δεν έχει περάσει και πολλή ε, χρόνος και πολύ πρόσφατα στη Νότια Κορέα. Και κάθε φορά είναι εκατοντάδε οι νεκροί. Γιατί έχουν πολλούς επιβάτες αυτά τα απορθμία και επίσης τα επιβατικά και επίσης βουλιάζουν και πάρα πολύ γρήγορα. Δέκα τροπολογίες, συγγνώμη 15 είχαμε εκτός από την έκθεση και συμφωνήσαμε να μην κάνουμε συμβιβαστικέ, αλλά να τις δούμε ξεχωριστά. Γιατί κάθε τροπολογία έβαζε το λιθαράκι της χωρίς να υπάρχει λόγος να τις ενώσουμε σε μια συμβιβαστική ή σε περισσότερες. Άρα είπαμε ότι συμβασμούς δεν κάνουμε. Στις τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε όλες ξεχωριστά. Λοιπόν, το βασικό μας θέμα ήταν να ορίσουμε τι είναι επιθεώρηση. Υπάρχει επιθεώρηση ε, ε, στο λιμάνι και επιθεώρηση εμπλό. Θα πρέπει αυτές να γίνονται ε, την ίδια χρονιά και να μην να μεσολαβούν πέντε μήνες τουλάχιστον ε, πρώτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα στις δύο αυτές επιθεωρήσεις. Να μην γίνεται δηλαδή τη μία μέρα πριν τον απόπλου του πλοίου και την άλλη μέρα εμπλό. Είπαμε πέντε με οκτώ μήνες για λόγους εκμετάλλευσης αφού το συζητήσαμε με διάφορους ενδιαφερομένους. Ε, δηλαδή και εκείνες που ναυλώνουν αυτά τα πλοία, οι τυφοπλιστέ, οι επιθεωρητές, είναι ο, ε, και τα πληρώματα. Επίσης ζητήσαμε στην έκθεσή μας να θεωρούνται πάντα ε, πλοία προτεραιότητα σε αυτά τα επιβατηγά σκάφη. Τα κράτη-μέλη είχαν κάποια διλήμματα και κάποια προβλήματα. Είτε δεν επιθεωρούσαν καθόλου αυτά τα σκάφη, είτε επιθεωρούσαν ορισμένα χωρίς να καλύπτουν την ποσόστοση. Αν χαρακτηριστούν σκάφη προτεραιότητας, ε, θα γίνονται σωστά οι έλεγχοι και επιθεωρήσεις και οι ποσοστώσει θα εξαντλούνται και η αιτήσια επιθεώρηση θα γίνεται, που είναι άλλωστε επιθυμητή. Επίσης έχουμε εισαγάγει και κριτήρια ε, υγείας και ασφάλειας του πληρώματος που δεν ε, προέβλεπε ο κανονισμό, για λόγους προφανείς για το πλήρωμα, αλλά και επειδή η ασφάλεια και η υγεία του πληρώματος έχει επιπτώσει και για τη γενικότερη ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών. Επίσης, αν αλλάξει χρήση η δρομολόγιο το πλοίο θα χρειάζονται νέες επιθεωρήσεις. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά υπάρχουν χώρες ε, που ζητούσαν να επαναληφθεί η επιθεώρηση. Όταν άλλαζαν δρομολόγια έτσι ώστε να βεβαιώνονται ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια. Πάντως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτά κυρία Πρόεδρε ε, είναι τα βασικά. Καλή συνεργασία, είχαμε καλό κλίμα ε, μπορεί να σα φαίνεται περίεργο, ε, συνήθω ότι δεν έχουμε συμβαστικέ, αλλά δεν ήθελε κανεί να έχουμε συμβαστικέ. Έχουμε λοιπόν σύνολο 28 τροπολογίε που θα τι ψηφίσουμε με τη σειρά. Και γενικά έχω θετικό πρόσημο στι τροπολογίες. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Η κυρία Μοντέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Ρικέ για τη δουλειά του και την όλη συζήτηση που είχαμε με θέμα αυτό το ντοσχέ. Σήμερα δεν έχουμε συμβαστικές λύσεις, διότι μπορέσαμε να υπερβούμε τις μικρές μας αποκλήσεις, ώστε οι τροπολογίες που αποβλήθηκαν να ικανοποιούν τους πάντες, όπως τις υπέβαλαν. Απλώς δύο μικρές παρατηρήσεις ως προς το θέμα, το ντοσχέ, την σημασία που δόθηκε στην ασφάλεια των σκαφών και το να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε όσο περισσότερο γίνεται τις τους διοικητικούς φραγμούς, τα διοικητικά άχθη. Για τις εταιρείε και την αλλαγή κατηγορίας. Εάν δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των σκαφών και εφόσον υπάρχουν επιθεωρήσεις συστηματικές, εδώ θα πρέπει να αφήνεται κάποια ευελιξία στην ε, έγκριση των αδειών, εφόσον έχουν ήδη ρυθμιστεί οι αρχικέ εκδόσει των αδειών. Ως προς τις επιθεωρήσεις υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες μπορούν να μην επιβάλλονται υποχρεωτικά. Εδώ πάλι για να μην έχουμε διπλές επιθεωρήσεις, διπλή χρήση των ίδιων πόρων και να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτήν την ανησυχία. Και μια τελευταία παρατήρηση, ο ορισμός του επιθεωρητού, επόπτη που θα πρέπει να καλύπτει και τους συγκεκριμένους επιθεωρητές από το κάτω σημαία και αυτούς του κάτω λιμένους. Θα πρέπει λοιπόν την τροπολογία που έχουμε υποβάλει και αντικατοτρίζει αυτήν την διάκριση για τους επιθεωρητές του κάτω σημαία να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει και αυτοί να έχουν την δυνατότητα να κάνουν τις επιθεωρήσεις. Και επίσης να φροντίσουμε η βάση των δεδομένων που θα δημιουργηθεί να καλύπτει και αυτή την κατηγορία σκαφών για να μην έχουμε πάλι διπλή χρήση των ίδιων συστημάτων. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Ρικέ και τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε την κυρία Ρικέ, ο κύριος Ουγελή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να Εδώ. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να συγχαρώ τον κύριο Ρικέ για την ε, συνεργασία μας στην έκθεση αυτή. Δεν το λέω μόνο ως σκιώδης εισηγητής, αλλά γιατί πραγματικά έχουμε συμφωνήσει στα περισσότερα θέματα, συμφωνώ και εγώ με τις περισσότερες λύσεις που έχουν βρεθεί Και όντω, σωστά ο εισηγητή εντόπισε σημεία που υπήρχαν επικαλύψει και επαναλήψει. Εδώ αναζητούμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Το σύστημα ελέγχων για τα οχηματαγωγά ρορό και τα ταχεία, ε, τα ταχαία, τα ταχύπλοα επιβατηγά πρέπει να γίνεται από τα κράτη-μέλη και με ένα σύστημα αξιολόγηση του κινδύνου. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, αλλά σε αυτό έτσι κι αλλιώ επικεντρώνεται η πρώτη μου τροπολογία. Θέλω, λοιπόν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ε, εκπροσωπήσω και την Ουγγαρία ως μια από τις μεγαλύτερες θαλασσίες δυνάμεις ε, παγκοσμίω. Αστείο ήταν αυτό. Ε, Απλώ προσπαθώ να μπω στην ίδια λογική με τα θελασσοπόρα έθνη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ουγγελή. Η κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα να πω. Ας προχωρήσουμε σε πλήρη συμφωνία. Κύριε Τέιλορ, εσείς τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Ε, πολύ καλή συνεργασία, επικοδομητικές συζητήσεις στις συναντήσεις των σκιωδών και στηρίζουμε πλέον στην έκθεσή σας. Η έκθεση είναι μάλιστα επίκαιρη, διότι θα γιορτάσουμε την 30η επέτειο από το επεισόδιο του, της Ζιμπρούγκε, της θάλασσας του Μπρούγκε. Ε, τότε που ένα φέρει δυστυχώς ε, προσέκρουσε και παρολίγο να βυθιστεί. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε όλα τα κράτη-μέλη ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ να αποφύγει οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν, ατυχέ συμβάν στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε λοιπόν για όσα κάνατε και θα σας στηρίξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω μόνο προς τον κύριο Ρικέ. Er ehm, ε, ε, υπάρχει ένα μνημόνιο ε, συνεννόησης των Παρισίων για την ασφάλεια τέτοιων σκαφών, εξ όσων γνωρίζω. Εμείς μετά όσα αποφασίζουμε στην Ευρώπη είμαστε στην ίδια κατεύθυνση με το εν λόγω μνημόνιο ή παίρνουμε έτσι δική μας ρότα και ακολουθούμε το ξεχωριστό μας δρόμο. Αυτή είναι μια ερώτηση γιατί υπάρχουν και θέματα διεθνούς ναυτιλίας και ναυσιπλοείας και κανόνες που τα διέπουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαντεγκάμπ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κοψένσκα. Είδατε έχουμε μια έκθεση που ζητάει διευκρίνηση για ορισμένα ε, θέματα και διατάξεις οδηγίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο επιθεωρήσεις. Και δανείζουμε τα λόγια των διαφόρων σχεδόν εισηγητών που χαρακτηρίζουν την έκθεση εξαιρετική. Και έχουμε και μια πρεμιέρα χωρίς τροπολογίες, συμβαστικές είναι αυτή η έκθεση. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, απαντήστε στις ερωτήσεις αυτές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ενώσω τη φωνή μου με όλων των υπολείπων συγχαίροντας τον κύριο Ρικέ. Ήταν ε, ιδιαίτερων τεχνικών λεπτομεριών αυτή η έκθεση και το όλο νομοθέτημα και όλες οι τροπολογίες αντικατοπτρίζουν την εξαιρετική δουλειά του εισηγητού. σε όλα αυτά τα στάδια. Καλωσορίζουμε τις τροπολογίες που διευκρινίζουν περαιτέρω αυτό που αυτή τη στιγμή συζητούμε. Και να απαντήσω αμέσω στην ερώτηση της Προέδρου για το ελάχιστο διάστημα μεταξύ των δύο ετήσιων θεωρήσεων, όπως είπε και ο κύριος Ρικέ, για να υπάρχει αρκετό χρόνο μεταξύ των θεωρήσεων είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δείξουμε κάποια ευελιξία για το ποια είναι καλύτερη στιγμή για να γίνονται επιθεωρήσει. Αυτό που πρότεινε ο κύριο Ρικέ μπορούμε να το δεχτούμε. Το δεύτερο σημείο που εγείρε ο κ. Ρικέ για κάποιες άλλες συγκεκριμένες τοπολογίες έχει να κάνει με το πώς συγκεκριμένα θα δούμε τα κάπως πιο επικίνδυνα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ το όλο επικίνδυνο. Δεν είναι ωραίο για τα ferry boat. Τέλος πάντων, για ένα σύστημα που θα μπορούσε να ε, ταυτιστεί με το σύστημα νιοψιών των λιμένων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι εθνικές αρχές. Οι λιμενικές αρχές σε πολλές περιπτώσεις. Αυτόν τον στόχο που επιδιώκεται, ίσως με μια νέα κάπως βελτιωμένη διατύπωση, και ε, αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 17, θα μπορούσαμε να βρούμε τη λύση. Και το επόμενο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ τώρα, είναι η τροπολογίες που καλωσορίζουμε πλήρως για την διευκρίνηση στην καθυστέρηση των υποβολών εκθέσεων ε, για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και την συμπερίληψή τους στην ε, βάση δεδομένων. Προβλέπονται 72 ώρες, ε, μάλλον προτείνονται 72 ώρες αντί για 24. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά την θέση της Επιτροπής Τραν και τους λόγους που έχει τέτοια στάση. Και τα ανέφερε και η κυρία Μοντέρο σε ό,τι αφορά την αλλαγή ε, κατηγορίας. Εδώ νομίζω ότι το θέμα που προσπαθείτε να καλύψετε με την τροπολογία σας ήδη καλύπτεται. Ίσως δεν είναι απολύτως απαραίτητο η τροπολογία αυτή να υπάρχει αλλά πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να το επιλύσουμε. Επίσης, κυρία Μοντέρο, αναφερθήκατε και στην επιστοποίηση και τα προσόντα των ε, επιθεωρητών. Συμφωνούμε ότι πρέπει να έχουν το κατάλληλο επίπεδο προσόντων. Να εξασφαλίζεται αυτό, διότι μόνο έτσι μπορούμε και εμείς να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας της επιθεωρήσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι σε κανένα σημείο διαφωνούμε προ τον επιδιωκόμενο σκοπό, λίγο ω προ το περιεχόμενο στη τύπωση τη έκθεση. Επίση, αναφερθήκατε στην ε, ανάγκη διασύνδεση των διαφορών βάσεων δεδομένων. Να εξηγήσω ότι αυτό που είχαμε προβλέψει εμεί, ότι η βάση δεδομένων για τα στοιχεία των επιθεωρήσεων θα βασίζεται και στην ε, βάση δεδομένων κοντά Τώρα το αν πρέπει να διασυνδέονται αυτές οι δύο βάσεις δεδομένων ή όχι είναι κάτι που αξίζει να το δούμε αργότερα και να το διευκρινίσουμε ενδεχομένω, γιατί δεν θα υπάρξει άμεση διασύνδεση των δύο συστημάτων επιθεωρήσεων. Όμως, όλες αυτές τις τροπολογίες, όπως και όλες τις ιδιαίτερες ανησυχίες σας και συγκεκριμένε πτυχές της έκθεσης, το λαμβάνουμε υπόψη γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλος της, ε, ολόκληρου του δικτύου των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και πάλι ο λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Ρικέ. Προσπαθώντα να απαντήσουμε ίσω και στην ερώτηση του κυρίου Βίντενκαμπ. Βάντενκαμπ. Παρακαλώ κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά θα απαντήσω. θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω τους αδέλφους ε, για τις παρατηρήσεις στα σχόλια και ιδιαίτερα για την ε, έγκριση και τη συνέλευσή τους. Σε σχέση με τα είπε η κυρία Μοντέρο για την αλλαγή δρομολογίων, την αλλαγή χρήση. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε μέρη στην παρατήρησή σας, που είναι πάρα πολύ εύλογη. Καλύπτεται όμως από το γεγονός ότι αυτό είναι δυνατότητα, δεν είναι υποχρέωση. Οπότε δεν θα επιβάλλουμε ούτε στο κράτος σημαία ούτε στο κράτος λιμένα κάτι το οποίο είναι δυνατότητα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να έχουν αυτή τη δυνατότητα, να κάνουν τις επιθεωρήσεις οι χώρες που το επιθυμούν. Δεν υποχρεώνουμε εκείνου που δεν το επιθυμούν, αλλά επιτρέπουμε σε εκείνου που επιθυμούν να διεξάγουν τι επιθεωρήσει αυτέ, γιατί αυτό ικανοποιούσε κάποια αιτήματα. Ξέρω, αυτό ήταν το μόνο θέμα ε, που είχαμε ε, συζητήσει με την κυρία Μοντέρο. Για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Βάντεν Κάμπ, βεβαίως δεν θα πάρουμε δρόμο ε, απέναντι ή αντίθετο με τις συμφωνίες των Παρισίων. Απλώς εμείς διευκρινίζουμε και προχωρούμε ε, πιο πέρα στον κανονισμό αλλά και στα παραρτήματα που είναι πιο σημαντικό συμπεριλαμβάνονται αυτές οι διατάξεις γιατί τα παραρτήματα ασχολούνται με τους τεχνικούς ορισμούς. Βεβαίως ευθυγραμμιζόμαστε και συμμορφωνόμαστε με το ε, μνημόνιο των Παρισίων. Δεν είμαστε ούτε εκτός ε, ούτε ε, απέναντι αλλά εντός του πλαισίου Ε, ακούσαμε επιφυλάξεις για την τροπολογία 17 που έχει να κάνει με τα παραρτήματα και ε, ε, επηρεάζει και άλλους κανονισμούς και άλλες νομοθεσίες. Ξέρετε ότι ε, πήγαμε να συναντήσουμε επιθεωρητές και μάλιστα εμπλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αιτήματα των κρατών μελών. Αντί να πούμε ότι ε, ενοχλεί που ενοχλεί η τροπολογία 17 και θα έχει και παράπλευρες επιπτώσεις και ε, πόλεις, αλλά ακριβώς αυτά τα σκάφη είναι σκάφη προτεραιότητας και τα δράματα και τραγωδίες και τα ναυάγια ε, ήταν πάρα πολύ ε, δαπανηρά και πρόκειται για πολύ νεκρά ναυάγια, για μεγάλες τραγωδίες. Είναι δυνατόν να τα παραγνωρίζουμε και να μην... Ας πούμε να ελέγχουμε φορτηγά τύπου 2 πριν τα φέρει μπότι, τα ρορό, γιατί στον κανονισμό τώρα είναι η σειρά του τάδε φορτηγού πλοίου και δεν μπορώ να κοιτάξω το επιβατηγό. Ε, κατανοώ αυτά που μας λέτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα συζητήσουμε στο τριμερή διάλογο να ακούσουμε το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη κατανοώ την ε, δυσκολία. Την έχουμε αντιληφθεί κι εμείς, αλλά προς το παρόν διατηρώ τη θέση μου αυτή, εκτός αν τα κράτη-μέλη αναθεωρήσουν. Νομίζω ότι ήταν ρήτη και ξεκάθαρη θέση τους. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλες οι τροπολογίες των συναδέλφων θα βελτιώσουν το κείμενο και τελικά θα έχουμε συνένεση και ευνοϊκό κλίμα και ευχάριστη διάθεση. Συνεχίζουμε με την ευχάριστη διάθεση, λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί την έκθεσή σας από τις 9 και μετά. Επόμενο θέμα, κανόνες και προδιαγραφές ασφαλείας για τα επιβατικά πλοία. Θα δώσω μέσα στο λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Αγιούτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε την τελευταία συνάντηση με τους κέντρους εισηγητές που επωφελούμε τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω διότι η συνεργασία μας ήταν πολύ επικοδομητική και γεμάτη από ιδέες και προτάσεις. Σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, προσπάθησα να καλύψω με αυτές κάποια από τα, σημαντικά, τα σημαντικότερα στοιχεία της πρότασης τροποποίησης της οδηγίας και κάποια σημεία που φαίνονταν κρισιμότερη σημασία από άλλα. Θα φαντάζεστε Ποιο είναι το πρόβλημα με το χάλιβα εδώ. Εδώ πρέπει να δούμε για τη Γαλλία τι θα ισχύει με το αλουμίνιο και την εξαίρεση που ζητάει. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές. Αρχές αυτές είναι ότι το αλουμίνιο είναι από τα υλικά που θα είναι ισοδύναμα. Εδώ δεν είναι το πρόβλημα το χαρακτηριστικό του ίδιου του υλικού, αλλά οι ιδιότητες του κατά πόσο ένα συγκεκριμένο μέταλλο μπορεί να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα με, με αυτά που προσφέρει. Έτσι καταλήξαμε στη συγκεκριμένη τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την ε, Γαλλία, το ισοδύναμο υλικό προβλέφθηκε έχοντας κατά νου ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της γαλλικής βιομηχανίας. Είναι ένα κράτος με ένα σημαντικό στόλο. Οπότε χρειάζεται κάποια περισσότερη ευελιξία. Για να είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούμε όσα προβλέπει η οδηγία. Γι' αυτό προβλέφθηκαν τα 8 συν 1 χρόνια σε ό,τι αφορά τη Γαλλία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας για να προχωρήσουμε στους τριμερείς διαλόγους με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που βρήκαμε τη δυνατότητα συμφωνίας με τους υπόλοιπους ε, εισηγητές είναι να βρούμε κατευθυντήριες γραμμές για τα σκάφη κάτω των 24 μέτρων. Βεβαίως ως προς αυτό ήδη έχει κάποια μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θέλουμε να προδικάσουμε ή να κάνουμε κι εμείς τα ίδια με αυτά που προβλέπουν τώρα στην Επιτροπή για τους διεθνείς κανόνες. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας σε καμία περίπτωση. Όμως, και όταν υποβλήθηκε το όλο θέμα στην κρίση μας, το θέμα ήταν, όπως είπαμε, να μην έχουμε γκρίζε ζώνες, ούτε νομοθετικά κενά. Δεν θέλαμε λοιπόν να παραγνωρίσουμε τους διεθνείς κανόνες ή να δημιουργήσουμε κρίζες ζώνες. Επίσης, η κατάσταση της Ελλάδας. Για την Ελλάδα καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία. Διότι εκεί όλα τα κράτη-μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει τον ορισμό των θαλάσσιων περιοχών και είναι σταθερά στη θέση τους. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η δυσκολία να οριστούν θαλάσσιες περιοχές αποκλειστικά και μόνο για την Ελλάδα, αντί για θαλάσσιες περιοχές θα μιλάμε για θαλάσσιες ρότες, θαλάσσιες πορείες. Είναι και αυτό μια κατάκτηση της οδηγίας. Τέλος, για την ε, βελτίωση της ασφάλειας ε, στη θάλασσα, και την ανάμειξη εδώ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να συνδυάσουμε την ασφάλεια με τα κοινωνικά θέματα και τι εργασιακέ συνθήκε. Θέματα που είναι αλληλένδετα και εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η ψηφοφορία θα γίνει λοιπόν αύριο. Γι' αυτό θα σας ζητούσα από, όλα τα, από όλες τις ομάδες να στηρίξετε την χρονοδότηση ε, αυτή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διακομματεύσεις με το Συμβούλιο και να μην χάσουμε τα υπόλοιπα σκέλη του νομοθετήματος του, της όλης μέτρων του Refit και να πάνε όλα αυτά ταυτόχρονα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γιούτο. Θα δώσω το λόγο τους, στους χιώδεις εισηγητές. Κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ συνοπτικός γιατί ειλικρινώ πρέπει να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. την ευαισθησία που έδειξε, καθότι η πρόταση της Επιτροπής πηγαίνει ακριβώς προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, την απλούστευση της οδηγίας, περιορίζοντας το κόστος και τους ελέγχους που ως τώρα δεν έχουν φέρει προς τη θέμενη αξία ως προς την ασφάλεια. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν πήγαινε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι με την ε, επιπλέον δουλειά της εισηγήτριας και όλους τους συναδέλφους Κιώδης, πετύχαμε ακόμη περισσότερο διάνα στο στόχο μας. Οπότε θα έχουμε ακόμη περισσότερη απλούστευση. Πέντε συμβαστικές τροπολογίες με τις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε και Εντό των προτάσεων αυτών καλύφθηκαν πάρα πολλέ άλλε τροπολογίε που είχαν ε, υποβάλει συνάδελφοι και από την ομάδα μου. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να εκφράσω την ειλικρινή ευχαριστία μου προ την εισηγήτρια. Και βεβαίω θα τη στηρίξουμε για τη διαπραγματευτική εντολή στου τριμερεί διαλόγου με το Συμβούλιο. Πιστεύουμε αύριο θα φανεί ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση από όλε τι ομάδε τη Επιτροπή μα. Για τους σοσιαλιστές, η Ιστιώδης η κυρία Γιάλα Σέντερ δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος που θα εκπροσωπήσει την ομάδα των σοσιαλιστών, κύριος Ερτούγκ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μόνο ένα ερώτημα. Γιατί μιλάμε. Για τη συνεργατική οικονομία ή όχι. Okay, sorry. Α, συγγνώμη, βιάστηκα. Θέλετε να πάτε πιο γρήγορα για το χρονόμετρο. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε, κύριε Αρτούκ, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στους ε, κανόνες και τα πρότυπα ασφαλής για την επιβατικά πλοία. Εκεί είμαστε, είχαμε ε, ολοκληρώσει τα ψηφιακά ζητήματα. Λοιπόν, η Αγιάλα Σέντερ δεν είναι εδώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Φώστερ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτριά μας και τις πολύ οικοδομητικές συναντήσεις που είχαμε. Νομίζω ότι ουσιαστικά οι περισσότερες σημαντικές προτάσεις είναι εντάξει, έχουμε εργαστεί πολύ αποτελεσματικά, ε, όμως υπάρχουν κάνα δύο θεματάκια που δεν μας βρίσκουν απόλυτα ικανοποιημένους. Το θέμα που αφορά τα βοηθητικά σκάφη, το πώς αντιμετωπίζονται από το Κοινοβούλιο, διότι το βοηθητικό σκάφος, η Λέμβος, είναι ουσιαστικά κάτι που αφορά τον εξοπλισμό του πλοίου. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε λοιπόν τη συμβαστική 2, διότι δεν είναι ένα πλοίο, πλοιάριο ε, αναψυχής αυτή η Λέμβος, αυτό το πεθητικό σκάφος και θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που λέμε. Έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες και κανονισμούς ε, και δεν θα ήταν σκόπιμο να έχουμε ένα ενωσιακό πρότυπο εφόσον έχουμε τα διεθνή πρότυπα που πρέπει να τηρούνται. Θα το θέσω και το είπα και στους σκιώδεις συζητητές. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί δεν είναι δεδειγμένο προς για τον κανονισμό αυτό. Σε ό,τι αφορά αυτά τα θαλάσσια δρομολόγια ε, που αναφέρουμε συγκεκριμένα την περίπτωση της ε, Ελλάδας, αυτό που ε, ήθελα να πω και ζήτησα και από τα σχέδια να το λάβει υπόψη είναι ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα μια χώρα που θα χρησιμοποιεί αυτά τα δρομολόγια αντί θαλάσσιες περιοχές ως σημείο αναφορά. Αλλά μπορεί γι' αυτό να ισχύσει και σε άλλες περιπτώσεις που θα χρειαστεί να προσωπικοποιηθεί αυτό ο διάδρομο, αυτή η περιοχή, αυτό, αυτή η ρότα. Ε, πρέπει να γραφτεί ξεκάθαρα. Ε, δηλαδή να αφήσουμε μια γενική αναφορά και να μην βάλουμε το όνομα της Ελλάδας, γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αυτό το θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε δει αντίστοιχε περιπτώσεις με νησιωτικέ περιοχές και άλλες χώρες. Γι' αυτό και το έχω ζητήσει. για την αύξηση των κοινωνικών προδιαγραφών και προτύπων για τους εργαζομένους. Φυσικά κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι το πεδίο εφαρμογής αυτό τη οδηγία συγκεκριμένη. Είναι η λάθο οδηγία, αν θέλετε, γιατί αυτό το τεχνικό έγγραφο βασίζεται στα πρότυπα τη σήμανση όλα. Ο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ε, Διεθνή Οργάνωση Εργασία. Δεν είμαστε δηλαδή ε, στο σωστό πεδίο εφαρμογής κατά την άποψή μου και σε ό,τι αφορά διασυνοριακές επιχειρήσει έρευνα και διάσωση. Εδώ μιλάμε για εσωτερικά δρομολόγια μόνο. Άρα πάλι είναι λάθος αυτή η αναφορά. Τέλος πάντων, συνολικά με αυτές τις ανησυχίες ε, και αυτά που λέω δεν είναι πολιτικά ζητήματα, έτσι είναι τεχνικά ζητήματα. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε, κατά τα λοιπά όπως είπα. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Απλά πρέπει να δούμε αυτά τα δύο-τρία ζητήματα πριν την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Foster. Madame Η κυρία Μπιλμπάου, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιούτο για την εργασία της. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στις πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες επί των οποίων συνεργαστήκαμε θα τις δεχτούμε και να πούμε ότι η συμβαστική 4 για το αλουμίνιο για το αν είναι ισοδύναμο ή όχι υλικό αυτό λύθηκε με τις διάφορες προθεσμίες που ετέθησαν για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και είναι ισόρροπη η λύση που βρέθηκε και λογική που μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγκληση στο μέλλον και συνένεση με την ε, λόγο ε, ρύθμιση. Αυτή είναι η θέση μας. Για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες ε, και τις πέντε συμβιβαστικές θέλω να τονίσω. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπιλμπάου. Κυρία Κίλωνεν, θέλει το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε. Πίτερ Βαντάλεν. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα να πω κάτι στους συναδέλφους για την αυριανή ψηφοφορία. Έχουμε μια τροπολογία υπαριθμών 39 δικιά μας. Μια τροπολογία κατά τα άλλα που ταυτίζεται με τη 40 του συναδέλφου Λούντγκρεν. Η η συγγητρία δεν θέλει να τις συμπεριλάβει στις συμβαστικές τροπολογίες. Εμείς θέλουμε όμως ε, να έχουμε ε, μια ε, ευθυγράμμιση του ορισμού των παραδοσιακών σκαφών με την Οδηγία 2295. Τα ιστιοπλοϊκά δεν συμπεριλαμβάνονται και επίση επικρατεί ασάφεια σε σχέση με τα παραδοσιακά πλοία. Προσέξτε, εδώ γίνεται λόγος για παραδοσιακά σκάφη επιβατηγά. Υπάρχουν όμως, Πρόεδρε, και κάποια παραδοσιακά σκάφη τα οποία ε, ποτέ δεν είχαν σχεδιαστεί ως επιβατηγά. Ε, ας πούμε, τα μεγάλα ρημουλκά ε, τα οποία τώρα όμως ε, ε, είναι εμπορικά και μεταφέρουν και επιβάτες, πάνω από 12 τα περισσότερα. Ε, δηλαδή, να βγει ο όρος επιβατηγά, η μεταφορά επιβατών, αλλά μιλήσουμε μόνο για παραδοσιακά ποντοπόρα πλοία. Δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί η συγγήτρια δεν το έχει συμπεριλάβει στην συμβαστική τροπολογία. Είναι κείμενη νομοθεσία Υπάρχουν μεγάλα ρημουρκά τα οποία τώρα έχουν αλλάξει χρήση και μεταφέρουν και επιβάτες εκτός από εμπορεύματα. Σας εφιστώ την προσοχή λοιπόν στις τροπολογίες 39 και 40. Στο τέλος θα απαντήσει η συγγήτρια και θέλω να ακούσω για ποιο λόγο δεν έχει συμπεριλάβει αυτές τις τροπολογίες μας στη συμβαστική. Τι την οδήγησε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ. Uh, uh, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να καλησπέρισω και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Γιούτο. Εξαιρετική δουλειά κυρία Γιούτο και η Σκιώδης το ίδιο. Πολύ επικοδομητικά και θετικά προσέγγισαν το θέμα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο της έκθεσης. Στηρίζουμε και τις πέντε συμβαστικές τροπολογίες αυτό που μας ικανοποιεί όμως ιδιαίτερος είναι η συμπερίληψη συμβιβαστική πρότασης για την κοινωνική διάσταση, για τους εργαζομένους όπου περιλαμβάνεται και η δική μου τροπολογία με την οποία τόνιζα πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε παρκή εκπαίδευση και κατάρτιση για το πλήρωμα ιδίω για τις επιχειρήσει τις διασυνορικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ευχαριστώ και περιμένω και εγώ την ψηφοφορία. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρικέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ το, την εισηγήτρια ε, και ως Γάλλος θα ε, μιλήσω και εγώ για το αλουμίνιο ε, και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια δεν θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να αντιμετωπίζονται έτσι τα πλοία από αλουμίνιο, δηλαδή ότι το αλουμίνιο είναι ισοδύναμο υλικό. Είναι τελείως ε, παράλογο αυτό. Ε, και νομίζω ότι χρειαζόταν ε, η προσπάθεια και πρέπει να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Το ζήτημα ε, βρέθηκε σε πολύπλοκη θέση η κυρία Γιούτο προσπαθώντας να χειριστεί κάτι που ήταν αδύνατο να χειριστεί γιατί η πρόταση ρύθμισης δεν ήταν η σωστή. Και συμφωνώ με αυτό που λέει ο κ. Βαντάλιν ε, για τα βατηγά πλοία και τα πλοία γενικώ. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την πρόταση της Κομισιόν που έβαλε και σε δύσκολη θέση το κοινοβούλιο και την εισηγήτρια. Ευχαριστώ την κυρία Γιούτο που έκανε ό,τι μπορούσε για ένα υλικό που δεν είναι ισοδύναμο, θα το κάνει ισοδύναμο, ε, και τέλο πάντων ε, το στρίβουμε από εδώ, το στρίβουμε από εκεί το θέμα, προσπαθώντα ότι θα καταλήξουμε στο τριμερή διάλογο σε μια διαπραγματευτική θέση και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αποδεκτή κοινή θέση. Τέλο πάντων, το πρόβλημα είναι η Κομισιόν με την πρότασή τη, ιδίω στα πλαίσια του Ρέφιτ. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητική αυτή η πρόταση. Θέλω να ευχαριστήσω πάντω την εισηγήτρια. Merci beaucoup, monsieur Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρικέ. Σε εσά ο λόγο και πάλι, κυρία. Ρεζένσκα για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των αγαπητών συναδέλφων. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα των εισηγητών που εργάστηκε για την οδηγία αυτή, ιδιαίτερα στην εισηγήτρια. Ήταν περίπλοκο, πολύ περίπλοκο το θέμα και από πολιτικής απόψεως, όπως γνωρίζετε, λεπτό και ευαίσθητο, ίσως περισσότερο από κάποια άλλα θέματα. Εμείς καλωσορίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνη που συνδέεται με τις μεταβατικές περιόδους για τα ε, σκάφη από αλουμίνιο. Ε, δράτω με τις ευκαιρίες αμέσως για να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Ρικέ ε, να επαναλάβω κάτι που είπα προηγουμένως. Αυτό βασίζεται σε διεθνή επιστημονικά στοιχεία που λένε ότι δεν είναι ισοδύναμο του ε, χάλιβα το αλουμίνιο, αλλά το αλουμίνιο με τη σωστή μόνωση μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο του χάλιβα. Και ακριβώς προς τα εκεί κατευθύνεται η οδηγία. Δηλαδή Έχουμε σκάφη ε, από αλουμίνιο και στο παρελθόν και σήμερα και στο μέλλον. Όποτε λοιπόν χτίζονται τέτοια καράβια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό η οδηγία αυτή να ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο θέμα. Και πάλι συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Είναι ισορροπημένος ο συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμέ, για σκάφη κάτω των 24 μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται αυτή τη στιγμή για ένα ε, κώδικα ε, μικρών σκαφών ε, για χρήση στα εθνικά χωρικά ύδατα και όχι στα διεθνή ύδατα. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή δρομολόγια ισχύουν τα διεθνή πρότυπα και κανόνες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια ε, που κάνει ε, διάκριση ανάμεσα στις θαλάσσιες ρότες, δρομολόγια και στις θαλάσσιες λεκάνες. Η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη γεωγραφική θέση και κατάσταση, όπου ε, ο όρος sea routes, οι θαλάσσιοι δρόμοι, τα δρομολόγια θα πρέπει να γίνει δεκτός. Για όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, αυτό μάλλον θα σημάνει ε, άχρηστη καθυστέρηση και ε, αναβολή της συμφωνίας. Επίσης, κάτι που ρώτησε η κυρία Φώστερ ε, για τις σωστικές λέμβους. Βεβαίως η λέμβη δεν είναι δεν είναι σκάφη αναψυχής. Ε, αλλά οι ε, διεθνείς κανόνες δεν ε, διέπουν τις λέμβους που μεταφέρουν τους επιβάτες από το πλοίο στην ξηρά. Και επίσης σε ό,τι αφορά την αλλαγή του πεδίου εφαρμογής που αποκλείονται παντός είδους παραδοσιακά σκάφη. Θέλω να σας πω το εξής. περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής εάν ε, κοιτάξουμε όλα τα παραδοσιακά σκάφη και μεταξύ αυτών εκεί ένα που έχουμε μετατραπεί σε επιβατηγά. Αυτό θα περιορίσει την εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχουν κάποια πλοία ε, που έχουν αλλάξει χρήση και έχουν γίνει επιβατηγά και κινδυνεύουν να μην υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ε, με τα όσα ορίζει η οδηγία. Ε, γι' αυτό, για τη συγκεκριμένη τροπολογία που ρωτήσατε. Και στη συγκεκριμένη οδηγία, όπως και στις δύο προηγούμενες, προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία μαζί σας για να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία και με τον άλλον συνομοθέτη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φώστερ. Θέλετε να επανέλθετε. Ευχαριστώ. Κάτι διευκρινιστικό θέλω να ρωτήσω. Για τις λέμβους λέτε λοιπόν. Βεβαίως, όταν χρησιμοποιούνται στα διεθνή ύδατα, καλύπτονται από τη σόλα στην αντίστοιχη σύμβαση. Αν χρησιμοποιούνται όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρια, χωρικά ύδατα ενός κράτους μέλους, είναι διαφορετική η κατάσταση. Λέτε ότι χρησιμοποιούνται για αναψυχή. Για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται για ψυχαγωγία, για, για περιήγηση. Όχι, συμφωνούσα ότι δεν χρησιμοποιούνται για αναψυχή και για τουρισμό. Αυτό εξηγούσα, ότι ε, τα διεθνή πρότυπα εφαρμόζονται μόνο όταν ε, χρησιμοποιούνται και στα διεθνή δρομολόγια. Ξέρω εγώ εκτός της Ενδεχομένω να μπορούν να χρησιμοποιούνται και εκτός ε, χωρικών υδάτων ενός κράτους μέλους. Οπότε εκεί ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί. Τουλάχιστον εγώ έτσι κατάλαβα τη δική σας παρέμβαση, ότι δεν κάνουν παράκτιο τουρισμό ε, οι Λέμβοι αυτές. Δεν ξέρω αν σας παρεξήγησα, παρανόησα όσα είπατε. Θα τα πούμε μετά το τέλος της συνεδρίασης διμερός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Of members of this committee. Πάντα είμαι στη διάθεση των μελών της Επιτροπής σας για οποιαδήποτε διμερή συνομιλία για να διευκρινίσουμε κάποιο θέμα. Μάλιστα. Καταλάβατε λοιπόν ότι είναι ανοιχτέ οι θύρε του γραφείου τη κυρία Κοσενσκά. Αν έχετε και άλλε ερωτήσει, γιατί εμεί θα συνεχίσουμε και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μα, την κυρία Γιούτο. Παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ συνάδελφοι για τη στήριξή σας. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις, ιδίως για την κυρία Φώστερ, τα ίδια μου είχε πει νομίζω και όταν συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα, στην τελευταία συνάντηση των Σκιωδών. Τα ίδια θα τις απαντήσω. Να υποφεληθώ για να απαντήσω και στον συνάδελφο Βαντάλεν σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 39 και 40. Τις στήριξα, απλώς δεν προέλεψα νέα συμβαστική, διότι για τον ίδιο παράγραφο, για το ίδιο δάφιο δεν υπήρχαν άλλες παρατηρήσεις ή τροπολογίες, οπότε δεν υπήρχε λόγος ή ανάγκη να προκύψει νέα συμβαστική. Αλλά στήριξη σίγουρα υπάρχει. Αυτά. Σας ευχαριστώ και ελπίζω αύριο ότι θα φανούμε ομόψυχοι. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Γιούτο. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί, από τις 9 και μετά. Και τώρα, πού πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε στην έκθεση κυρίας Κίλονεν. Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο της Εργατική Οικονομία, κυρία Κίλονεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί ήσασταν ιδιαίτερο δραστήριοι και είχατε πολύ θετική ε, προσέγγιση απέναντι στη συνεργατική οικονομία. Είχαμε 152 τροπολογίες στην νομοδότηση και μπορεί ως ε, πολιτικό να μην είναι πολύ ιδιαίτερα ικανοποιημένη και ω δηλαδή πρέπει να το πω μετά από δύο συναντήσει ε, με του Σκιώδη νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας για τη συνεργατική οικονομία, νομίζω ότι είναι θετική συνολικά. Ιδίω ό,τι αφορά του τομεί ε, του τουρισμού και των μεταφορών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο κλάδος των μεταφορών, ο κλάδος του τουρισμού δημιουργούν πολλές θέσει εργασίας βάσει της συνεργατική οικονομίας και προσφέρουν προσιτέ τιμέ και εναλλακτικέ υπηρεσίες. Επίσης, δημιουργούν νέες ε, δυνατότητες, νέες εισοδηματικές πηγές ε, προσφέρουν και δημιουργούν και ένα νέο πλαίσιο ε, ρύθμισης των υπηρεσιών αυτών. Μπορούμε να έχουμε ένα ευφυές νέο πλαίσιο που θα προωθεί την καινοτομία και τους στόχους πολιτικής της Ένωσης, παραδείγματος χάρη περιορισμό των εκπομπών άνθρακα, πρόσβασιμότητα των μεταφορών και παροχή περισσότερο σε προσιτές τιμές. Θέλαμε να προτείνουμε διατάξεις ε, που θα διευκολύνουν τις εξελίξεις. Η Κομισιόν πρέπει να παρακολουθεί την αγορά, να την ε, αναλύει ε, διεξοδικώς και εφόσον χρειαστεί να λαμβάνει δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή να μην δίνουμε φάρμακο στον ασθενή πριν αρρωστήσει, αλλά αφού αρρωστήσει. Πρέπει πάντως η υλοποίηση της ομοθεσίας να γίνεται με μεγαλύτερη επιμέλεια. Και οι φορείς της αγοράς θα πρέπει να έχουν ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού σε τα φορά και τις κοινωνικές συνθήκες για να υπάρχει ένα δίκαιο περιβάλλον ανταγωνισμού sinne, missä voitot syntyvät. Θα πρέπει επίση οι φόροι και τα άλλα τέλη, να καταβάλλονται στο χώρο, στον τόπο τη οικονομική δραστηριότητα. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία και τα μέσα για να μπορεί να γίνεται αυτό. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πολύ επιτυχημένα, από την Εστονία για παράδειγμα, τα οποία θέλουν να ε, βρουν μιμητές και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την παρεκονομία και τη φοροαποφυγή. Έτσι θα γίνει πιο αποδεκτή η εργατική οικονομία. Θα ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι προδραστική στην προσέγγιση της. Και καλό και όλα τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τους φορείς της συνεργατικής οικονομίας μεταξύ των ε, ε, πλεκομένων φορέων τους οποίους έχουν επαφές και διαβουλεύσεις. Ελπίζω όταν ρυθμιστεί ε, με την ατζάντα αυτή η συνεργατική οικονομία να βασίζεται στο γενικό, σε γενικούς τομεακούς κανόνες. Δεν νομίζω ότι βιώσιμη λύση θα ήταν να υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την συνεργατική οικονομία. Έχουν γερθεί κάποια ερωτήματα, κάποια ερωτηματικά σε σχέση με την επιρροή τη συναλλακτική οικονομία στην αγορά εργασία. Εμεί θα θέλαμε πάντω να υιοθετήσουμε στην Επιτροπή μα μια θετική προσέγγιση, τονίζοντα ότι η αγορά εργασία μεταβάλλεται και πω η συνεργατική οικονομία μπορεί να προσφέρει δυνατότητε, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίε. για τα άτομα τα οποία μέχρι τώρα δυσκολεύονταν να βρουν τη θέση του στην αγορά εργασία. Παρ' όλα αυτά, καλούμε την Επιτροπή να επαγρυπνά και να βλέπει κατά πόσον τα κοινωνικά και ασφαλιστικά συστήματα των κρατών μελών προσαρμόζονται ε, στις νέες μορφές εργασίας του πλαίσιο της εργατικής οικονομίας. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας ε, και σε κάποιες δραστηριότητες ε, επιμερισμού, κόστος επιμερισμού κερδών Υπάρχουν και κάτι άλλοι όροι, car sharing, car pooling, αυτός ο λεγόμενος συνεπιβατισμός. Όλα αυτά έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές ε, στην αγορά εργασίας και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει τις ε, διαφορές. Τότε ό,τι το σύστημα μεταφορών, τα συνεργατικά οικονομικά μοντέλα νομίζω ότι μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συγκοινωνικών ε, μοντέλων, να μειώσουν ε, τις εκπομπές, τις συμφορήσεις και έτσι να αξιοποιηθεί το δυναμικό αυτό. Βέβαια για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουμε ολοκλήρωση των παραδοσιακών συστημάτων και των νέων ε, συστημάτων ε, συνεργατικής οικονομίας. Πρέπει να υπάρχει διαπαφή, πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να προωθούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες ή άλλες πρωτοβουλίες που θα αφήνουν εκτός ε, του σχεδιασμού, των μεταφορών κτλ. τη συνεργατική οικονομία. Τα συστήματά μας δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά και θα πρέπει να υποστηρίζονται οι επιβάτες, οι χρήστες των ε, συγκοινωνιών και των μεταφορών σε όλη την ε, αλυσίδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη θετική συμβολή και προσέγγιση τους και ελπίζω βέβαια ότι θα υποστηριχθούν και συμβαστικές προτάσεις αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κίλονεν. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μοντέρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Κιλόνεν για την ε, λεπτομερέστατη αυτή παρουσίαση, αλλά και τόσο σφαιρική σε σχέση με την έκθεση αυτή. Πράγματι, φτάσαμε να έχουμε μια έκθεση πολύ θετική σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε αρχικά στα πλαίσια της συνεργατικής οικονομίας και αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε είναι να διευκρινίσουμε λίγο την νομοθεσία και να θεσπίσουμε νομοθεσία που ήδη βέβαια υπάρχει αλλά πιο απλουστευμένη με αρχές που να δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές, κάποιους γενικούς προσανατολισμούς ώστε να υπάρχει συνέπεια και ορθότητα στους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε φραγμούς στις νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, γιατί υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη διάσταση που αφορά και τις μεταφορές και τον τουρισμό και θα πρέπει αυτές τις εναλλακτικές λύσεις που διαρκώς προκύπτουν ε, προς όφελος των καταναλωτών ή των επιχειρήσεων να μην τις εμποδίζουμε. Η συνεργατική οικονομία επίσης τονώνει το επιχειρήν, το πνεύμα του επιχειρήν. Επίσης, μια παρατηρήση για τα όσα έγιναν από την Γενική Διεύθυνση Growth για την προσαρμογή σύντομη διάρκεια, τη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή. Εδώ και στην ε, τροπολογία 47 έχουμε μία ανάγκη προσαρμογής των επαγγελματικών ενώσεων και των ομοτήμων. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίζει να υπάρχει κατάλληλη δουλειά στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας χωρίς να δημιουργούνται φραγμοί αλλά διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τους πολίτες με ε, ισότιμους κανόνες και να υπάρχει και ένα σωστό ε, κλίμα ανταγωνισμού ώστε αυτές οι νέες μορφές δημιουργούν κατανεμητικές ε, μορφές δραστηριότητας που πρέπει όμω να εφαρμόζονται με την απαραίτητη ισότητα και δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μοντέρο. Κυρία Ερτούκ, εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη κυρία Ταπαρντέλ γιατί έχει συνεδράσει στο Βουκουρέστι. Οπότε με χαρά να παρουσιάσω τις δικές της θέσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Ταπαρντέλ βεβαίως θέλει να συγχαρεί πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για την ε, καλή δουλειά της και την ισορροπημένη κυρίως προσέγγιση που επέλεξε. Η συνεργατική οικονομία είναι ένα νέο συναρπαστικό φαινόμενο, αλλά χρειάζεται με προσοχή να το ρυθμίσουμε για να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο υποστηρίζει το τελικό κείμενο της έκθεση κυρία Ταπαρντέλ που καταλήγει ότι είναι πολλά τα ωφέλη για την οικονομία από τη συνεργατική οικονομία αλλά έχει και κάποια χαρακτηριστικά προβληματικά. Για τον κλάδο των μεταφορών η συνεργατική οικονομία μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα ιδιαίτερα από τη σκοπιά της καλύτερης χρήσης υφισταμένων δυνατοτήτων και να έχει πρόσβαση στις λιγότερο προσβάσιμες περιοχές. Για τον τουρισμό επίσης έχει αυξηθεί και διαπορροφηθεί η προσφορά ε, και ανταποκρίνεται αυτό στην αυξημένη ζήτηση των τουριστών. Θα πρέπει όμως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική διάσταση και το κατά πόσο ευελιξία και ευκαιρία στην εργασία δεν συνοδεύονται με επισφαλείς και κακοπληρωμένες δουλειές. Χρειάζεται βαθιά ανάλυση λοιπόν για τις ε, προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με τη φορολόγηση και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία της φορολόγησης ε, των ε, εταιριών εκεί που παράγεται το κέρδος τα επιχειρηματικά μοντέλα του μέλλοντος είναι εκείνα τα οποία φορολογούνται ε, με δικαιοσύνη ε, στον τόπο που παράγουν κέρδη. Η συνεργατική οικονομία αλλάζει με γρήγορους ρεγδαίους ρυθμούς, έχει διαφορές ανάμεσα σε διάφορα κράτη-μέλη και φορείς. Παρ' όλα αυτά η ομάδα μας, στους πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα νέα μοντέλα θα πρέπει να ε, συνεργαστούν για να βρουν με ποιο τρόπο σωστά θα συμμορφωθούν και με καλή θέληση πάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρτούκ. Κύριε Ντάλτον, καλή σας μέρα. Μου χαμογελάτε και μου αρέσει αυτό. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Bonjour. Merci beaucoup, Madame President. Ah. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Η ιδιαίτερη εισηγήτρια ήταν πάρα πολύ πρόθυμη να δεχτεί τι προτάσει μα και είναι και πολύ καλέ ε, προτάσει. Υπάρχουν μερικοί τομεί όμω που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε του συμβιβασμού Πρώτον, δεν συμφωνούμε με την ανάγκη να εναρμονιστεί ε, σε ένα πλαίσιο. Είναι κορσές αυτό. Η οικονομία συνεργατική διαφέρει πάρα πολύ από κλάδο σε κλάδο και θα πρέπει να είναι ε, τομεακή η ρύθμιση, όχι εναρμονισμένη. Επίσης το παρα τραβάει η γνωμοδότηση για την αγορά εργασία. Η συνεργατική οικονομία είναι θετική για εργασιακά δικαιώματα. Έχουν ευελιξία οι εργαζόμενοι που δεν είχαν στο παρελθόν. Δεν είναι ε, σκλάβοι ενός αφεντικού ε, που τους ορίζει πόσες μέρες ε, άδεια θα έχουν και πότε θα λείπουν. Είσαι ίσα αυτό χειραφετεί τους εργαζομένους και δεν το αναγνωρίζει η γνωμοδότηση ως τα όφιλε. Επίσης δεν συμφωνούμε με την παραδοχή ότι το πρόβλημα είναι η συνεργατική οικονομία ε, για την φορολογία ή δεν μπορούμε να τη στιγματίζουμε έτσι. Και όπως είπε ο σοσιαλιστής συνάδελφος, γενικά υπάρχει πρόβλημα στη φορολόγηση, δηλαδή να φορολογούνται εταιρείε εκεί που παράγουν το κέρδος, αλλά αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα. Και το γενικότερο πρόβλημα των πολυεθνικών, όχι μόνο της συνεργατικής οικονομίας. Και πολλοί ε, ε, όπως είναι η Uber δεν πληρώνουν κέρδη διότι δεν έχουν, δεν πληρώνουν φόρο συγγνώμη γιατί δεν παράγεται κέρδος. Ε, προσοχή να μην είμαστε υπερβολικά αρνητικοί. Και αυτό το βασικό πρόβλημα που έχω με την έκθεση θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο θετικοί απέναντι στην εργατική οικονομία. Ε, είναι πραγματικά κάτι που δίνει δυνατότητες στον τουρισμό και στις μεταφορές ε, στον καταναλωτή. Εκεί ανθεί πραγματικά και οι επιβάτες είναι πλέον καταναλωτές. και αν είναι κακή η υπηρεσία που παρέχει στην εργατική οικονομία, αλλάζει πάροχο. Σηκώνεται και φεύγει ο καταναλωτή, ο τουρίστα, ο επιβάτη. Ε, σε σχέση με κάποιε παραδοσιακέ ε, προσφορέ ε, υπηρεσιών. Και είναι καλό και για το περιβάλλον. Δηλαδή όταν έχουμε συνεπιβατισμό σε κάποια αυτοκίνητα που διατίθεται για, κοινό έτσι, για κοινή χρήση, ε, είναι και καλό για το περιβάλλον και κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα στις πόλεις. Γενικά υποστηρίζουμε την έκθεση, αλλά με κάποιες συμβιβαστικέ έχουμε προβλήματα και το ύφο και η προσέγγιση είναι γενικά πολύ αρνητική για ένα τομέα που για μας είναι ιδιαίτερα θετικός και στο μέλλον θα βοηθήσει πολύ και τον τουρισμό και τις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάλτον, ο κύριος Καταρχάς ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Κίλωνεν. Έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Βλέπουμε ότι διαφέρουν οι απόψεις για τη συνεργατική οικονομία. Ε, υπάρχει μια στάση που είναι προοδραστική και θεωρεί ότι τα θετικά θα πρέπει να τα υπερτονίσουμε και μάλλον προς τα εκεί το σκέφτομαι κι εγώ και μια άλλη τάση είναι πιο δύσπιστη, πιο καχύποπτη και λέει ότι υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να ε, αναδειχθούν. Πάντα αυτό συμβαίνει με αναδυόμενα μοντέλα. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, υπάρχουν τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι. Ορισμένοι επιμένουν στα πλεονεκτήματα και άλλοι ε, στα μειονεκτήματα. Και όταν κάποιο έχει την άποψη, διαφωνεί με εκείνον που, που επιμένει στη βήτα. Η κυρία Κίλον προσπάθησε να βρει τη χρυσή τομή και τη το αναγνωρίζω. Η έκθεσή τη ε, συνάδει με την ε, έκθεση που είχα ε, παρουσιάσει εγώ και ενέκρινε η Επιτροπή μα ένα παρόμοιο θέμα, παρεμφέρει πριν από λίγε εβδομάδε. Δεν έχει περάσει πολλή χρόνο και ήταν σημαντικό να έχουμε κάποια συνέπεια, γιατί θα ήταν κάπω ενοχλητικό να είναι τόσο αποκλίνουσες οι εκθέσεις μας. Γενικά η πολιτική μου ομάδα θα στηρίξει τις προτάσεις που έχουν γίνει, αλλά συμβιβασμοί είναι αυτοί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, του συμβιβασμού, ότι δεν ικανοποιεί πλήρως τους πάντες. Δεν είναι ούτε όλα άσπρα, ούτε όλα μαύρα, κύριε Ντάλτον. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Η συνεργατική οικονομία έχει ε, βοηθήσει την ε, ασφάλεια στην παροχή υπηρεσιών, δηλαδή είναι πιο ε, κοντά ο πάροχος με εκείνον που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, γνωρίζεται ο πελάτης με τον πολιτή ας πούμε και υπάρχει πιο άμεση σχέση. Υπάρχουν επίσης κάποιες περιφέρειες στην Ήπεθρο που δεν έχουν μόνιμες συνδέσεις ε, για μόνιμα δρομολόγια. Δεν ξέρω, μπορεί να μην συμφωνώ, πάντα με εξέπληξε λίγο αυτή η αναφορά. Γενικά δεν έχω πάρα πολλά σχόλια. Μπορεί να θέλαμε ένα πολύ πιο αισιόδοξο τόνο, έτσι και πολεμοχαρή ε, και χαρούμενο, αλλά το είπε και ο Ισμαήλ Ερτούκ, ότι θα πρέπει να αναβάνουμε υπόψη και τις εντάσεις που υπάρχουν και ε, τα προβλήματα και τους φόβους και τις αγωνίες ορισμένων. Γενικά στηρίζουμε την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ρικέ. Είχα γράψει και εγώ το όνομά μου ως κυριώδης ε, εισηγήτρια. Κυρία Κίλωνεν, σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική σας ε, εργασία εδώ στη συγκεκριμένη νομοδότηση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η έκθεση. Το πρώτο μήνυμα της έκθεσης αυτής είναι ότι η συνεργατική οικονομία Χρειάζεται οπωσδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο και εδώ στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας λείπει αυτό. Αυτό το ρυθμιστικό προθεσμικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί από τη μια θα πρέπει να έχουμε ορίσει το περίγραμμα αυτής της δραστηριότητας που δεν ορίζεται με σαφή τρόπο ε, και υπάρχουν κάποιες ε, καιροσκοπικές ε, πλατφόρμες Όλες οι πλατφόρμες αυτές δεν είναι της συνεργατικής οικονομίας, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι ε, φορείς συνεργατικής οικονομίας που είναι πλατφόρμες. Εγώ δεν θέλω ψευδεπίγραφες τέτοιες πλατφόρμες. Η συνεργατική οικονομία έχει να κάνει με κάτι που μοιράζονται οι χρήστες. Και απευθύνομαι στον κύριο Ντάλτον που μας έδωσε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα και μας μιλάει για την εταιρεία Uber. Κύριε Ντάλτον, η Uber είναι μια υπηρεσία μεταφορών που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη πλατφόρμα ως διεπαφή. Και αυτή ε, είναι παροχή υπηρεσίας επαγγελματική, εξού και η διαφορά που πρέπει να έχουμε ανάμεσα στη συνεργατική οικονομία και την ε, οικονομία ε, όπου οι πολίτες μοιράζονται διάφορα πράγματα και υπηρεσίες. Η συνεργατική οικονομία θα πρέπει να παραμείνει σε παροχή υπηρεσιών μη επαγγελματικών, για να μην έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό σε παραδοσιακές εμπορικές παροχές, ταξί, λεωφορεία κτλ. Υπάρχει κίνδυνος κοινωνικού ντάμπινγκ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση κυρίως αυτοαπασχολούμενοι είναι εκείνοι που παρέχουν την υπηρεσία και δεν έχουν συγκλίνει ακόμα οι κανόνες για τις κοινωνικές εισφορές και ε, τα λοιπά ε, ε, καθήκοντά του. Ας μην είμαστε αφελεί. Δεν πρόκειται κανείς να αποφύγει την επαγγελματική χρήση τέτοιων πλατφόρμων, διότι η νεολαία είναι δυναμική και η τεχνολογική επανάσταση είναι γεγονός δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα ε, σε σχέση με τις τεχνολογίες εξελίξεις. Ερωτώ λοιπόν, τι γίνεται με αυτές τις ε, πλατφόρμες, πολλαπλασιάζονται και είναι επαγγελματικές επαναλαμβάνω και πώς το αντιμετωπίζουμε. Πρώτον, προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει μια οροφή ε, στο εισόδημα ή να φορολογούνται από ένα όριο και μετά και το όριο να αναφέρεται σε κάθε κλάδο χωριστά ή σε κάθε πλατφόρμα ή θα μπορούσαμε να φανταστούμε και ενιαίο για όλες τις συνεργατικές δραστηριότητες. Όλα αυτά δεν τα εξτάζει έκθεση, δεν αποφαίνεται οριστικά, χρειάζεται ουσιαστική ευρωπαϊκή νομοθεσία και εδώ ε, σκέφτομαι και την έκθεση του κυρίου Ρικέ που είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Η Επιτροπή Μεταφορών περιλαμβάνει τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Ε, όταν κανείς μοιράζεται αυτοκίνητο, ας πούμε, ε, και άλλες, αλλά εγώ ζητώ μια ξεχωριστή προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τουρισμό και για τις μεταφορές, όπου το θεμελιώδες ερώτημα και ζήτημα είναι η προστασία των καταναλωτών ή προστασία των ε, δεδομένων και περιμένω να δώσετε συνέχεια. Και θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου, κυρία Κίλωνεν, ότι η έκθεση αυτή δεν θα πρέπει να παραμένει στα σερτάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει έρθει η ώρα να μας δώσει πραγματική λύση για αυτά τα προβλήματα, που τώρα μόλις αναδύονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Λοιπόν, τα είπα Ελπίζω να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά συνεχίζουμε τους και ηγητές. Ο κύριος Ντεμές Μάκερ, παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι σκιώδης ηγητής, αλλά να μιλήσω. Είχα ζητήσει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κίλωνεν και τους ε, σκιώδης ηγητές. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και έχω, έχω κάνει κάποιες ε, τροπολογίες και χαίρομαι που βλέπω ότι εγκρίθηκαν και έχουν συμπεριληφθεί ε, στις συμβαστικές της εισηγήτριας. Άρα για μένα είναι ξεκαθαρό ότι η συνεργατική οικονομία ε, μπορεί να φροντίσει για τις μεταφορές και τον τουρισμό να ανθεί στην Ευρώπη. Έχει πλέον εκτήματα για τον καταναλωτή, για τον περιβάλλον και για τις επιχειρήσεις Συμφωνώ πολύ με εκείνους που λένε ότι υπάρχουν γκρίζε ζώνες και κατακαιρματισμός στην νομοθεσία που θα πρέπει να καλυφθούν και να ε, αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, κοιτάξτε, θα πρέπει να φροντίσουμε η συνεργατική οικονομία να μην ε, έχει μια προσέγγιση από πλευρά μας πάρα πολύ άκαμπτη. Έχει ένα χαρακτήρα ευέλικτο και αυτορυθμιστικό και αυτά απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση. Η νέα νομοθεσία λοιπόν θα πρέπει να βασίζεται σε βαθιά ανάλυση, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαίτερότητε των διαφόρων κλάδων τη συνεργατική οικονομίας. Ασφάλεια δικαίου, αναλογικότητα και ε, προσεκτική αντιμετώπιση θα πρέπει να πριτανεύουν. Άρα, συνάδελφοι, είναι και δικός μας ρόλος να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό κλίμα για ε, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αξίζει να ενισχυθεί αυτή η οικονομία για να είναι ισχυρή και να ευδοκιμήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Δεμόντε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες ή λιγότερες φιλοδοξίες, αλλά πετύχαμε να είμαστε θετικοί στην προσέγγιση μας. Και είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες πτυχέ, διότι η εναλλακτική είναι να έχουμε ένα κατακαιρματισμένο ή ενίο και συνεπές πλαίσιο. Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει κάθε κράτο το δικό του νομοθετικό σύστημα και του δικού του κανόνε. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε εδώ στην Ευρώπη, είναι ένα αναγνωρισμένο πλαίσιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραβλέψουμε και τις, ε, τα επιτεύγματα που έχουμε πετύχει ως τώρα. Έχουμε, θέλουμε να έχουμε θεμετό ανταγωνισμό, νόμιμο και θεμητό ανταγωνισμό. Θέλουμε να έχουμε την ίδια φορολογία για όσου προσφέρουν τι ίδιε επαγγελματικέ υπηρεσίε, αλλά να προσφέρουμε και τα ίδια πρότυπα ασφάλεια. Διότι η ασφάλεια είναι ήδη κάτι που, αποτέλεσε επίτευγμα για του παραδοσιακού τομεί. Θέλουμε να το αποτύχουμε αυτό λοιπόν με την νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και με τι κυρώσει οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές ε, επιπτώσεις στο τι επιλέγετε. Επηρεάζεται έτσι και ο Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγητρία που έλαβε υπόψη και την ανάγκη η φορητότητα των δεδομένων, η δυνατότητα μεταφοράς τους δηλαδή να λαμβάνεται υπόψη ακόμα και από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή διαλλακτικότητα και ευελιξία. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε, ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια. Έχω καταθέσει ορισμένε τροπολογίε ε, που συμπεριλαμβάνονται στις συμβαστικέ τροπολογίε, και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γι' αυτό. Το θέμα είναι σίγουρα η μείωση τη χωρή, η μείωση των εκπομπών, αλλά και οι θέσει εργασία, ε, ε, οι οποίε όμω θα πρέπει να έχουν μια κοινωνική διάσταση και να είναι ενθαρρυντικέ. και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ θετικό επίση που δίνεται σημασία στην κινητικότητα πρέπει και στην Ήπεθρο να εξασφαλιστεί κινητικότητα χωρίς ε, να χρειάζεται να βασιζόμαστε πάντοτε στο αυτοκίνητο. Μια άλλη παρατήρηση, λίγο πιο αναλυτική, το είπε και ένας προλαλή σας, ε, ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι σκλάβοι. Και εγώ θα έλεγα δεν πρέπει να είναι σκλάβοι οι εργαζόμενοι. Και εμείς ε, ε, το φροντίζουμε αυτό με τους ε, οδηγούς φορτηγών για παράδειγμα. Είχαμε έναν Ρουμάνο οδηγό που στην Γερμανία και στην Ολλανδία οδηγούσε ένα φορτηγό για 8 μήνες και κοιμότανε το βράδυ εκεί. Δεν μπορούσε να πάει καν σπίτι του. Και έπαιρνε νομίζω γύρω στα 250 ευρώ ε, μισθό. Αυτό είναι πραγματικά μοντέρνα δουλειά, μοντέρνα σκλαβιά. Και αυτό πραγματικά πρέπει να το πούμε. Ε, υπάρχουν άλλοι, είμαστε σε άλλε εποχέ τώρα και όλα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται. Αν δεν ελέγχονται, δεν χρειάζεται να έχουμε και την σχετική νομοθεσία. Ε, αυτή ήταν η μία παρατήρηση. Δεύτερη, ευελιξία. Ότι θα πρέπει επιχειρήσει, επιχειρηματικέ να είναι ευελικτέ πράγματι και θα πρέπει να έχουμε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο. Θετικά όλα αυτά. Αλλά η καινοτομία σε ποια κατεύθυνση πηγαίνει. Για παράδειγμα, το, ε, για παράδειγμα πριν από δύο-τρει εβδομάδε στην ARD είχαμε για τη Ryanair μία ταινία και είδαμε πώ ε, αντιμετωπίζουν και πώ πληρώνουν του πιλότου στη Ryanair, η οποία είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεν έχουν ε, ασφάλεια, δεν, του δεν τους πληρώνουν φόρους. Δεν είναι αυτή η καινοτομία, η ευέλικτη, πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση και θα πρέπει να φροντίσουμε. Φυσικά και θέλουμε να έχουμε ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες και αν δεν είναι κοινωνικά σωστές, τότε ε, δεν είναι σωστός και ο ανταγωνισμός. Και η Κομισιόν έχει το ρόλο να τα προσέχει όλα αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά αφορά τους πιλότους της Ryanair. Εδώ και 10 χρόνια υπάρχουν ε, προβλήματα, ε, υπάρχουν ε, όλες αυτές οι επιφυλάξεις. Τα ξέρει η Κομισιόν και δεν αντιδράει εδώ και 10 χρόνια. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μας πει η Κομισιόν τι κάνετε εσείς σκέφτεστε συγκεκριμένη αυτή περίπτωση της Ryanair. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι ε, κερδίζουν και ωφελούνται από όλα αυτά είναι αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν την νομοθεσία και χρησιμοποιούν τους σύγχρονους εργαζόμενους ως σκλάβους. Merci, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Κύριε Νίλσον. Ευχαριστώ. Εδώ σήμερα συζητούμε τη συνεργατική οικονομία. Στη Σουηδία πρέπει να σας πω ότι Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, νέες δυνατότητες. Ε, πολλές μέθοδοι μάλιστα είναι πραγματικά σαρπαστικές. Από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε και προβλήματα. Δεν υπάρχει μόνο θετική πλευρά, υπάρχει και αρνητική. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν πολλοί να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα ε, στο πλαίσιο της εργατικής οικονομίας, στον τομέα των μεταφορών, που θα μπορούσε εκεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά βέβαια και πάντα υπάρχουν μικρές εταιρείε, μεταφορικές εταιρείε. Πάντα υπήρχαν, για παράδειγμα, σε διάφορους τομείς προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε για να έχουμε οικονομίες και έχει λειτουργήσει θετικά. Είναι ένα συνεργατικό μοντέλο, ε, ουσιαστικά μοντέλο συνεργατικής οικονομίας που ισχύει εδώ και καιρό. Δηλαδή μην λέμε συνέχεια ότι είναι ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Μην είναι λίγο κουραστικό αυτό, γιατί υπάρχει εδώ και καιρό. Και η συγγήτρια είπε ότι υπάρχει πράγματι κίνδυνο ε, να υπάρξει φόρο αποφυγή. Υπάρχουν συμβουλευτικέ εταιρείε για παράδειγμα, σήμερα που συμβουλεύουν επιχειρήσεις και λένε ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα με τα οποία μπορείτε να εξοικονομήσετε ε, από φόρους ε, ή να μην ικανοποιήσετε κάποιες, ε, κάποιους όρους, κάποιες απαιτήσει σε ό,τι αφορά την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων εργασιακών. Και αυτό είναι ελκυστικό για κάποιες επιχειρήσεις. Υπάρχει λοιπόν ε, αυτό ο κίνδυνος, αυτά τα νέα προσφέρουν επιχειρηματικά μοντέλα και νομίζω ότι θα πρέπει να, είμαστε, να επαγρυπνούμε απέναντι σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίλσεν. Βίρκουνεν, παρακαλώ κύριε, μέχρι το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ καλή συνεργασία μας με, με την εισηγήτρια, διότι κατάφερε να συνδυάσει πολλές διαφορετικές ιδέες σε συμβαστικές λύσεις για το θέμα της συνεργατικής οικονομίας. Προφανώς δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο μόνο για, όλα τα, για όλες τις προεκτάσεις της συνεργατικής οικονομίας. Προφανώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και κλάδοι ε, είναι διαφορετικό δηλαδή το πώ ενοικιάζονται διαμερίσματα ή πώ προσφέρονται υπηρεσίε εστίαση ή τι γίνεται με τι υπηρεσίε μεταφορών. Δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να τα καλύψουμε με ένα και μόνο νομοθέτημα. Σε κάθε κράτο μέλο, προ στιγμή, έχουμε πολύ διαφορετικέ συνθήκε για το πώ μπορεί κανεί λόγου χάρη να νοικιάσει ή να μισθώσει προσωρινά ένα διαμέρισμα. Οπότε, Υπάρχουν κάποια στοιχεία της συνεργατική οικονομίας που θα πάρουν άλλη κατεύθυνση από ό,τι κάποια άλλα. Βεβαίω ο σκοπός είναι, είτε βρισκόμαστε στο διαδίκτυο είτε όχι, είτε, παροχή είτε μιλάμε για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών είτε όχι, να είναι μια παράλληλη πραγματικότητα αυτή που διαμορφώνονται. Τώρα είναι πολύ διαφορετικέ οι νομοθεσίε των κρατών μελών, όπω βλέπουμε σε πολλά σημεία. Λόγω χάρη για το Uber. Έχουν τελείω διαφορετική νομοθεσία για το θέμα των ταξί, των ε, οχημάτων που μισθώνονται για σύντομε μεταφορέ τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη για να είναι νόμιμος ανταγωνισμό και να μην επιβάλλονται ίδιε υποχρεώσει στους διάφορους κλάδους. Δεν μπορεί δηλαδή να προκύπτουν νέε υπηρεσίε και νέοι κλάδοι που να μην έχουν καμία νομοθετική ρύθμιση και κάποιοι άλλοι να είναι επιβαρημένοι. Πάντω, είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει αυτέ τι κατευθυντήριε γραμμέ, βασιζόμενοι στο γεγονό ότι τα κράτη-μέλη θα δώσουν περισσότερο χώρο στι νέε εταιρείε. Διότι έχουμε επενδύσει εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη για την διασύνδεση στο ίντερνετ και έτσι έχει προχωρήσει και η ηλεκτρονική παραχή υπηρεσιών. Δημιουργούνται διαρκώ νέε υπηρεσίε, νέε μορφέ υπηρεσιών. Βλέπουμε οι καταναλωτέ να τι θέλουν, να τι επιζητούν. Είναι πολύ δημοφιλεί. Οπότε θα πρέπει να αφήσουμε και κάποια σχετική ελευθερία στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν του κανόνε του όπω θέλουν και να υπάρχει και ένα περιθώριο για κοινοτομία. Να ξαναπώ ότι δεν πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό ότι θα έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο και μόνο για ολόκληρο το ε, ζήτημα της ε, συνεργατικής οικονομίας. Κυρία Βίρκουνεν, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα στρέφω το βλέμμα μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την κυρία Βανχάνεν από, την από τη Γενική Διευθύνση Grow, Βανχάνεν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που πήραν αυτό το λόγο. Η συζήτηση ήταν ε, πρόσφορη και μας έδωσε πολλές χρήσιμες ιδέες. Όπως πολλοί βουλευτές σημείωσαν σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ ήταν να τονίσει ότι πιστεύει. Πιστεύει ότι υπάρχει πολύ δυναμικό και πολύ δυνατότητα ανάπτυξη στην εργατική οικονομία και θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση με τόσο γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης θα πρέπει να προσαρμόσουμε αναλόγως και την νομοθεσία μας. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, διευκρινίσουμε τους κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προβλέψουν τους δικούς τους ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι εταιρείες θα έχουν την ίδια μεταχείριση, το ίδιο σημείο αφετηρίας όταν παρέχουν υπηρεσίες. Και κυρίως όταν παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Βεβαίω και για του ιδιώτε, αλλά και στην περίπτωση των αξιολόγηση ομοτήμων, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κάποια όρια τηρούνται ώστε να διαχωρίζονται και οι επαγγελματίες από τους απλούς ιδιώτε. Όπως παρατήρησαν πολλοί βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να μελετά τον τομέα αυτό και έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον τουρισμό και τις παροχές υπηρεσιών υποδοχής επισκεπτών. Εκεί η Επιτροπή μελετά τον κλάδο αυτό γιατί ε, εξελίσσεται γοργά και με διάφορες μελέτες που έχουμε βλέπουμε οι οποίες θα διατεθούν μέσα στο 2017, βλέπουμε πώς μπορούμε να εκφράσουμε καλύτερες προτάσεις σε πολιτικές που να συνδυάζονται και με τη συνεργατική οικονομία. Θα συνεχίσουμε βεβαίως να είμαστε σε επιφυλακή, ώστε να ισχύουν οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί κανόνες μεν και να εφαρμόζονται και σωστά στα επιμέρους κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν άκουσα το λόγο. Ο λόγος μάλλον είναι ότι σήμερα έχετε τη διάθεση να διακρίνετε σαφώ τα πράγματα, όπως είπατε και προηγουμένω. δηλαδή επαγγελματικέ υπηρεσίε από τη μια με όσα αυτό υποκρύπτει και επιφέρει. Δηλαδή δραστηριότητα επαγγελματική πολύ καλά πλαισιωμένη και η συνεργατική οικονομία. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβω σήμερα είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βλέπει ότι το θέμα αυτό πραγματικά είναι όλο και πιο δημοφιλές και έχει μεγαλύτερη διάδοση και δημιουργική προβλήματα στα κάτι Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποφασίζει επιτέλους να σκεφτεί ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο διότι αναφέρθηκε από διάφορους βουλευτές εδώ. Γιατί κάποια στιγμή να μην φτάσετε να πείτε έχουμε ένα θέμα το οποίο διαρκώς και περισσότερο είναι διαδεδομένο και θα προλάβουμε λίγο τις εξελίξεις. Δηλαδή να μην να βρούμε κάποια νομοθετική βίωδο διότι όταν μιλάμε για συνεργατική οικονομία και δεν κάνουμε καμία διάκριση, και τα αφήσουμε να εξελιχθεί αυτό ανεξέλεγκτα, μετά όταν θα πάμε πίσω να αποκαταστήσουμε τι βλάβε, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να προλάβουμε λίγο. Η πρόνοια είναι καλύτερη από την θεραπεία. Γιατί να μην κάνουμε κάτι με νομοθετικού δρόμου και διόδου, ώστε να πλαισιώσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή. Όταν ε, συνέτασε αυτή την ε, ε, ανακοίνωση για την συνεργατική οικονομία είχε υπόψη ότι αλλάζει ραγδαία, ότι νέα επιχειρηματικά μοντέλα αναδύονται, παλιά εξαφανίζονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να βρει κάτι που να ε, ισχύει για όλους τους κλάδους της οικονομίας αυτής. Άρα θεωρήσαμε ότι ήταν πρόωρο ακόμα το στάδιο. Τη στιγμή που εγκρίθηκε η ε, ανακοίνωση για την συνεργατική οικονομία. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επιχειρηματική οικονομία, ε, αυτή η συνεργατική μάλλον, πώς θα είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα και από εκεί και πέρα θα ε, αντιδράσουμε. Χρειάζεται να γίνει μια διαβούλευση, να ολοκληρωθεί, γιατί διεξάγεται αυτό το καιρό και βλέποντας και κάνοντας. Έχω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Είναι η οικονομία του αύριο αυτή. Και εγώ δεν θέλω η Επιτροπή Μεταφορών μας να ε, είναι δακτυλοδεικτούμενοι ότι δεν θέτουμε τις σωστές ερωτήσεις. Όλοι οι συνάδελφοι έκαναν πολύ καλές ερωτήσεις. Και τι μας λέτε προς το παρόν δεν κάνουμε τίποτα γιατί δεν μπορούμε να τη φρενάρουμε αυτή την οικονομία. Πείτε μου όμως σήμερα, ε, ε, τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις μεταλέτες τις έχετε στα σερτάρια σας. Η κυρία Βίρκουνεν σας έκανε πολύ καλή ερώτηση προηγουμένως. Είπατε ότι θα πρέπει να κάνετε μια αξιολόγηση. Μελέτες έχετε. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές. Μετά εμείς ε, ως Επιτροπή Μεταφορών θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Πού βρίσκεστε λοιπόν. Όπως σας είπα προηγουμένως κυρία Πρόεδρε, πολλές γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγουν διάφορες μελέτες ή το έκαναν στο παρελθόν για τη συνεργατική οικονομία. Ξέρετε ότι όταν αναθέτει μια μελέτη χρειάζεται πολύ χρόνο να έρθει το αποτέλεσμα, να δημοσιευθεί, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Μόλις ολοκληρώνεται το κάθε θέμα, εμείς ε, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των μελετών. Κατά τη διάρκεια του λοιπόν, θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα καλύψουμε και τον τομέα των μεταφορών. Δηλαδή μόλις ε, θα τι έχουμε στα χέρια μα θα διατεθούν, θα δημοσιοποιηθούν. Κύριε Κράμερ πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, μα εγώ έκανα και μια ερώτηση που δεν απαντήσατε όμω. Εγώ είπα ότι τα δύο τρίτα των πιλότων στη Ryanair δεν έχουν σωστή σχέση απασχόληση. Εδώ και 8 χρόνια το ψάχνετε. Αποτέλεσμα δεν βγάζετε, όλο το ερευνάτε. Ούτε ναι δεν μα λέτε, ούτε όχι. Για, τι κάνετε και γιατί αδρανείτε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ε, Mm, uh, uh, Ο λόγος για τον οποίο δεν έθιξα αυτό το θέμα στην απάντησή μου είναι ότι δεν έχει άμεση σχέση αυτό με τη συνεργατική οικονομία, το θέμα της εργοδότησης των κυβερνητών οι μελέτες που κάνουμε εμείς περιορίζονται στη συνεργατική οικονομία και μόνο. Euh, Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούμε. Η συγγήτρια, η κυρία Κίλωνεν, παρακαλώ να κλείσει. Αύριο ψηφίζουμε από τις 9 και μετά. Vous avez la Voilà, la parole est Εντάξει, ακούτε. Ωραία. Μπορείτε να ολοκληρώσετε ως ε, καθελήν αρμόδιο Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω από καρδιάς όλοι να αναγνώσετε τις συμβαστικέ λύσεις που συντάξαμε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές ώστε να καταλάβουν όλοι ότι η υπομονή ανταμείβεται. Βλέπουμε ότι παρά τις διάφορες δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζονται πρέπει να δείξουμε υπομονή και παρά τις διάφορες καθυστερήσεις θα χρειαστεί αργά ή γρήγορα η προσέγγιση της ενιαίας αγοράς των διασυνοριακές υπηρεσίες βλέπουμε να ε, είναι όλο και περισσότερο διαδεδομένες. Εδώ χρειάζεται δηλαδή μια προσέγγιση ε, ενιαίου πλαισίου με συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλιώς θα καταλήξουμε να είμαστε σαν τα παιδάκια που παίζουν στην παιδική χαρά σε έναν αμόλοφο και κάποια στιγμή κλειστράνε, σαν σε τσουλήθρα. Θέλουμε λοιπόν έναν τομέα ο οποίος να είναι κάπως ελεγχόμενος παρόλο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ελπίζουμε να έχουμε και τις κατόλληλες μελέτες με τα διάφορα στοιχεία ανάλυσης και με τρόπο ώστε να περνάνε καλύτερες πρακτικές από το ένα κάτω μέλος στο άλλο. Να αξιοποιούνται αυτές οι καλύτερες πρακτικές και να μην επαναλαμβάνουμε λάθη που έχουν διαπραχθεί και αλλού. Κατά την άποψή μου, Πρέπει όλοι να ε, ηρεμήσουμε κάπως, να πάρουμε κάποια απόσταση από το θέμα για να το δούμε αντικειμενικά, αλλά να μην είμαστε και υπερβολικοί και αδρανίσουμε, να είμαστε διαρκώς επιφυλακοί για την συνεργατική οικονομία συνολικά. Και να πω στον συνάδελφο, τον κύριο Ντάλτον, ότι είμαι από τη Φιλανδία και συγκεκριμένα από μία επαρχία έναν νομό όπου οργανώνονται ιδιαίτεροι, όπου μάλλον το καλοκαίρι μας κάνει να είμαστε ιδιαίτεροι, ιδιαίτερα απεσιόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ αποτιμώ να είμαι αισιόδοξη, ό,τι και αν συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. σοφορία ε, της έκθεσης αυτής θα ψηφιστεί όπως και οι υπόλοιπε εκθέσεις αύριο από τις 9. Να συνεχίσουμε τώρα με την πρόταση για την προώθηση της διασύνδεσης στο ίντερνετ των τοπικών κοινοτήτων. Ο λόγος στον κύριο Ερτούγκ, διότι η κυρία Ταπαρδέλ δεν μπορεί να έρθει. Και ζητά συγγνώμη. Ε, ο κύριος Ερτούγκ, ευχαριστώ πρόεδρε. Και πάλι θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος κυρίας Ταπαρδέλ και να παρουσιάσω τη θέση της για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Συνάδελφοι, η διασύνδεση στο διαδίκτυο είναι σύνδεση μάλλον, προϋπόθεση και προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να λειτουργεί σωστά η οικονομία. Θα πρέπει να είναι δωρεάν, ασφαλές ε, και εύκολο στη ε, πρόσβαση. Wi-Fi for EU λέγεται αυτό και ε, προσπαθεί να δημιουργήσει μια λειτουργούσα ενιαία ψηφιακή αγορά δίνοντας ελεύθερη σύνδεση σε δημόσιους χώρους παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εισηγήτρια λοιπόν η κυρία Δαπαρτέλη είχε ένα διπλό στόχο. Πρώτον, να εξασφαλίσει ότι το δωρεάν ε, ασύρματο διαδίκτυο θα αφορά και τις τουριστικές τοποθεσίες και ε, τις υπηρεσίες μεταφορών. Αυτό μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να βελτιώσουν ε, τις τουριστικές οδούς και να βελτιώσουν και τη ζωή των πολιτών. Αντίστοιχα, για τον τουρισμό Όταν ε, υπάρχει το διαδίκτυο είναι πιο ελκυστικοί οι προορισμοί και οι τοποθεσίε. Συμφώνησαν όμω ε, οι ε, στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή είναι περιορισμένοι οι πόροι που διατίθενται, ότι μπορεί η πρωτοβουλία αυτή να θεωρηθεί ε, ως μία κίνηση δημοσίων σχέσεων. Ε, θα πρέπει να δοθεί σωστή προβολή για να μάθουν οι πολίτες την πρωτοβουλία αυτή και οι δήμοι και οι κοινότητες. Να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει και θετικά για τους πολίτες, για την καθημερινή ζωή τους και αυτό ε, θα πιάσει τόπο και αν γίνει με συνετό τρόπο. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε πέρα από τις δημόσιες σχέσεις και να προσπαθήσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειάζονται επενδύσεις και εδώ θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξη όλων των συναδέλφων για τις τροπολογίες που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει την πρικοδότηση της συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η ποιότητα χρειάζεται και απαιτεί σοβαρές επενδύσεις. Σε σχέση με αυτό, κάτι που τονίσαμε όλοι στις διαπραγματεύσεις ήταν σημασία να έχουμε μια σωστή γεωγραφική ισορροπία ε, στα σπότ αυτά του ασύρματου διαδικτύου. Θα πρέπει να δημιουργούνται εκεί που χρειάζονται περισσότερο σε όλα τα κράτη-μέλη και ε, σε αστικές και σε υπαίθριες περιοχές. Και επίσης ε, επιπλέον χρηματική υποστήριξη είναι κάτι το κρονού κάνευ. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι συμβατό το πρόγραμμα με κάποια άλλα περιφερειακά ε, προγράμματα ή κρατικά ή ας πούμε το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και να έχουμε συνέργειες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ερτούκ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βίρκουνεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ζήτρα και τους κοιόδης εισηγητές. Είναι μάλλον πολύ σημαντικό να έχουμε γρήγορες συνδέσεις ε, και τεχνολογίε πληροφοριών επικοινωνιών σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ καλό για τι υπηρεσίε για του πολίτε και η πρόταση αυτή αφορά την προώθηση καλύτερων συνδέσεων, ασύρματων συνδέσεων στους κοινόχρηστους χώρους, δημόσιους χώρους. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε πολλές περιοχές έχουμε ήδη ε, γρήγορες ε, διαδικτυακές συνδέσεις βάσει αγοράς. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες επένδυσαν στις συνδέσεις αυτές σε πολλές περιοχές στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι η βασική γραμμή και στο μέλλον. Για να βελτιώσουμε λοιπόν τη συνδεσιμότητα, πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι ο δίκαιος και αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι καλό να δημιουργούμε υποχρεώσεις ε, εκεί που ήδη είναι καλή η σύνδεση μπορεί να έχει ε, γίνει με κινητά δεδομένα ή με ασύρματη τεχνολογία. Σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται τα κινητά δεδομένα σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό δεν υπάρχει ασύρματη ε, συνδεσιμότητα τόσο πολύ. Δεν υπάρχει τόσο πολύ Wi-Fi. Βέβαια είναι σημαντικό τώρα να προωθήσουμε και τις επενδύσεις στις περιοχές που δεν είναι τόσο γρήγορες οι συνδέσεις ιδίως στους δημόσιους χώρους. Για τους, οποίες, ε, για τους οποίους αναφέρεται, στους οποίους αναφέρεται αυτή η πρόταση. Σημειώσαμε αυτό που είπε η ότι δηλαδή θέλουμε καλύτερες, καλύτερες συνδέσεις εκεί που υπάρχουν ε, κόμβοι εφοδιαστικής ή μπορεί να είναι τουριστικές περιοχές και οι δημόσιες συγκοινωνίες επίσης να έχουν ασύρματο δίκτυο. Ε, αυτά είναι τα βασικά που ενδιαφέρουν εμάς στην Επιτροπή Μεταφορών. Θέλω να ευχαριστήσω και, τις χιώδεις, και τους συγητές για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε κυρία Βίρκουνεν. Ευχαριστώ Σονέσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας γιατί είχαμε πολύ καλή συνεργασία, εργαστήκαμε επικοδομητικά και την κατάρτιση και των συμβαστικών προτάσεων. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένε πτυχές που είναι κάπως προβληματικές για το μέλλον κατά την άποψή μου. Εύρος του προγράμματος. Έτσι όπως προβλέπετε και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι τα δοχεία και οι πόροι που διατίθενται ετησίως, νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μήπως το μέλλον αλλάξει το πεδίο εφαρμογή και δεν θα ξέρουμε τι να υποστηρίξουμε, τι προγράμματα να υποστηρίξουμε. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις δημόσιες συγκοινωνίες και στους τουριστικούς χώρους. Και καλό είναι στις τουριστικές περιοχές να καλύψουμε συγκεκριμένα, συγκεκριμένους συγκοινωνιακούς κόμβους. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ένα δωρεάν δίκτυο. Αυτό θα επηρεάσει τον τουρισμό και τον συντονισμό της τοπικής κοινωνίας της πόλης, της εκάστοτε. Πρέπει να δούμε επίσης την οργάνωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Μήπως επηρεαστεί τιμή του εισιτηρίου, για παράδειγμα. Αυτό είναι άλλος τομέας. Δεν έχει να κάνει με την ε, συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. με βάση τους διαθέσιμους πόρους δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πράξει τεράστιος αντίκτυπος στη συμβα... συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ουσιαστικά είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που θα δίνει κίνητρα και θα επιτρέψει να βελτιωθεί σε τοπικό επίπεδο η συνδεσιμότητα. Και με επίκεντρο, όπως είπα, τουριστικές περιοχές και σε δημόσιες συγκοινωνίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο προπολογισμό. Η αύξηση του προπολογισμού μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί δεν είναι σαφές τι θα γίνει σε αυτό το πρόγραμμα, τι πόροι μπορεί να διατεθούν για την αύξηση αυτού του προϋπολογισμού. Και σε ό,τι αφορά τους όρου χρήση. θα πρέπει και εδώ τα οικονομικά θέματα να ρυθμιστούν για να μην υπάρξει ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα. Το είπε και συνάδελφος. Ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι στα ταχύτητα συνδεσιμότητας, αλλά να δοθεί βοήθεια σε διάφορους χώρους ή σε ιδιωτικού φορείς. Επίσης ούτε η ποιότητα της σύνδεσης είναι το μόνο κριτήριο. Εφόσον μπορεί τους νέους χώρους να ανταλλάσσονται τεράστιο και δεδομένων. Η αύξηση της ταχύτητας λοιπόν ίσως να μην είναι απαραίτητη πάντοτε. θα συζητήσουμε ε, με τους κοιοδησηγητές. Έχουν ληφθεί νομίζω υπόψη παρατηρήσεις μου. Θέλω να ευχαριστήσω μια ακόμη φορά την εισηγήτρια και τους συναδέλφους μου, τους κοιοδησηγητές και ελπίζω οι συμβαστικές αυτές προτάσεις να υπερψηφιστούν γιατί θα δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε βελτίωση της συνδεσιμότητάς σα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Λε Πρόεδρο. Συνεχίζουμε. Ο Ζάτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ε, τη συνάδελφο για τις συμβαστικές τροπολογίες και τις συζητήσεις που είχαμε. Η πρόταση αυτή είναι αρκετά μετριοπαθής ε, αλλά δεν έχουμε αρκετή εικόνα για το τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Ε, ποιοι θεσμοί είναι αυτοί στους οποίους ε, απευθυνόμαστε. Με τις τροπολογίες μας προσπαθήσαμε να διευρύνουμε τον αριθμό των θεσμών και να δούμε πού θέλουμε να έχουμε γρήγορο ίντερνετ. Επαναλαμβάνω, αυτή η πρόταση είναι μετριοπαθής, δεν είναι υπερβολικά φιλόδοξη και πρέπει να είναι πολύ καλά στοχευμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε κάθε φορά όταν προτείνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες μέχρι που φτάνει το χέρι μας. Ε, πάντως να δούμε ένα πρώτο αποτέλεσμα αυτή τη πρωτοβουλία όσο μετριοπαθής και αν είναι και όσο περιορισμένα τα χρήματα και ε, πώς θα γίνει χρηματοδότηση από 50 σε 120 εκατομμύρια δεν το βλέπω πάρα πολύ ε, πιθανό. Ε, στις τελευταίες συμβιβαστικές τροπολογίες, στη τελευταία έκδοση τους, γίνεται λόγος για δημόσιες μεταφορές, δωρεάν δημόσιες μεταφορές. Αυτό είναι μια είναι προβληματική από μόνη της, διότι έχει να κάνει με την αρμοδιότητα των ε, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συχνά είναι δημοτικές οι συγκοινωνίες και δεν μπορούμε να εξασφαλίζουμε παντού ε, συγκοινωνίες δημόσιες. Αυτό είναι θέμα επικουρικότητας και αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Θα πρέπει λοιπόν να ε, μιλάμε για τις αστικές συγκοινωνίες τουλάχιστον. Ε, οι αστικές συγκοινωνίες όμως δεν είναι κάτι το, εμπίπ, το οποίο εμπίπτει στη σημερινή συζήτηση. Γι' αυτό η ομάδα των φιλελευθέρων έχει πρόβλημα. Στη συνέχεια, συμβαστικές τροπολογίες 5 και 6 δεν γίνεται λόγος για τα νησιά. Γίνεται λόγος για περιφέρειες που εμφανίζουν κάποια οικονομική υστέρηση. Αλλά στην αρχική εκδοχή γινόταν λόγος για τα νησιά, τα οποία έχουν εξαφανιστεί στην τελευταία πρόταση που είδαμε λίγο νωρίτερα, πριν από λίγες ώρες. Για ποιο λόγο? δεν αναφέρονται όταν μιλάμε για περιοχές της Υπέθρου, Ορεινές και άλλες. Για ποιο λόγο έχουν εξαφανιστεί τα νησιά από αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθει και να διατηρηθούν. Γιατί όταν απαριθμούμε όλες αυτές τις περιφέρειες, καλό θα ήταν για λόγους ισορροπίας να παραμείνουν όλες οι ε, περιφέρειες αυτές. Ευχαριστώ, κυρία Εύαντς. Thank you, Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, την εισηγητρία. Νομίζω ήταν πολύ καλή συνεργασία μας για το θέμα. Ήταν ε, μια μακρά διαδικασία. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε και να προωθήσουμε την διασύνδεση στο ε, διαδίκτυο σε όλες τις περιοχές, ιδίως τις περιοχές της υπαίθρου. Είμαι βέβαιο ότι σε όλα τα κατημέλια υπάρχει κάτι παρόμοιο. και να πω ότι στη δική μου τη ομάδα, όταν είδαμε την αρχική πρόταση της Επιτροπής, και όπως ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της εισηγητρίας, ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια όμως μπορούμε να στηρίξουμε τι συμβαστικέ ε, τροπολογίες με την εξαίρεση μία της 12 Η Η τροπολογία που συμπεριλαμβάνει την ε, παράταση του σχέδιου κατά τρία χρόνια, του προγράμματος κατά τρία χρόνια και εδώ έχω βάλει σχετική τροπολογία που αναφέρεται όχι μόνο στη διάρκεια του ίδιου του προγράμματος, αλλά και στο ποσό που θα πρέπει να προβλέπετε. Ε, ήταν διαφιλονικούμενο το ποσό με το οποίο θα πρέπει να πληκοδοτηθεί το πρόγραμμα αυτό. Ε, εγώ και η ομάδα μου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον προϋπολογισμό και να χρησιμοποιηθεί από τα μη δαπανηθέντα ποσά του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε ε, να μην αφιερώσουμε υπερβολικά μεγάλα ποσά πριν δούμε τα πρώτα και επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Εύανς. Κυρία Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια και τους Κιώδης. Και παίρνω το λόγο για να τονίσω και εγώ από πλευράς μου την ανάγκη να Υπάρχει κάλυψη ίντερνετ σε όλες τις τυπικέ κοινότητες. Όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις και είναι αυτές που περισσότερο προστατεύονται αλλά και στι περιοχέ τη Υπέθρου, τι απόκεντρε και τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η σύνδεση στο ίντερνετ θα πρέπει να θεωρείται ω δημόσια υπηρεσία. Ω τέτοια υπηρεσία λοιπόν δεν μπορεί να, να είναι κάτι που επιφυλάσσουμε μόνο σε συγκεκριμένα μέρη της επικράτειας. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει την ίδια πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μια όθηση. Υπάρχει μια τάση αστιφιλίας. Οι περισσότερες, περισσότερα απομακρυσμένες περιοχές γνωρίζουν την απερίμωση, την εγκατάλειψη μάλλον από τους κατοίκους τους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε τις ανάλογες υπηρεσίε όπως θα κάναμε και για τις μεταφορές. Γι' αυτό έχω υποβάλει σχετικά τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω μια άλλη πτυχή. Δηλαδή ότι υπάρχει το δικαίωμα ε, πληροφορίας. Το δικαίωμα πληροφορίας που ακολουθεί τις τάσεις της ψηφιοποίησης ακόμα και στο επίπεδο της δημοσιογραφία με τις ανάλογες αλλαγές στις τιμές. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης στον στο διαδίκτυο με χαμηλές τιμές και δωρεάν, στο Wi-Fi. Αλλά και ο τουρισμός είναι ένας κλάδος που επηρεάζεται εδώ και είναι μια ζωτική σημασία σε υπηρεσία που ε, επιβάλλει την εύκολη διασύνδεση στο ίντερνετ και την απαιτούν και οι δύο καταναλωτές. Ευχαριστούμε κυρία ο κύριο Στελίντσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσυπογράφω στην ε, θέση των υπόλοιπων ε, σκιωδών εισηγητών από τους φιλελεύθερους αλλά να κάνω και εγώ δύο-τρία σχόλια. Πρώτον, κατά την άποψή μου, το πρόγραμμα αυτό δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις εθνικές προσπάθειες, δραστηριότητες και πολιτικές ή προγράμματα κατά την άποψή μου, είναι ένα κερασάκι στην τούρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώνει κάπως αυτά που ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνονται. Καταλαβαίνω πάντως ότι σε κάποιες χώρες είναι πιο ριζωμένες αυτές οι συνήθειες, σε κάποιες άλλες όχι. Εδώ θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει διασύνδεση στο Wi-Fi, στο διαδίκτυο, σε όλα τα κατημέρια και σε όλες τις περιοχές τους. Είναι δύσκολο βέβαια να υπάρξει ένα μόνο ενίο πρόγραμμα και καταλαβαίνω αυτό που είπε η κυρία Evans για τη διάρκεια, την παράταση. Σίγουρα θα θέλαμε περισσότερη διάρκεια για την τήρηση του ελέγχου από τις αρχές, τρία χρόνια, όμως το πρόγραμμα ε, προβλέπει μια σωστή μετάβαση και έχουμε τριπλασιάσει και τους πόρους του προγράμματος. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, ναι υπάρχουν και δημόσιες μεταφορές, είμαστε Επιτροπή Μεταφορών, αλλά είναι τελείως διαφορετικό το θέμα των μεταφορών. Μιλάμε για το πώς θα επηρεαστούν οι εγκαταστάσεις, οι κόμβοι, ε, το υλικό που χρησιμοποιείται στις μεταφορές, αλλά είναι διαφορετικά τα μέσα μεταφοράς. Εδώ ε, ο τρόπος που αναπτύσσονται είναι τελείως διαφορετικός. Αυτό βέβαια ήταν κάποια μελλοντικά σχόλια που καταφέραμε να έχουμε στο νου μας και στο μέλλον, γιατί φαντάζομαι ότι σε καμιά διετία θα, έρχεται, θα έρθει κάποιο να πει να λήξει το πρόγραμμα σε δύο χρόνια και θα ήταν κρίμα, θα κρίμα να διακοπεί απλώ και να έχει αποτύχει όλη αυτή η πρωτοβουλία. Θα πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία στα ίδια τα κράτη-μέλη για να γίνει σωστά η προσαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Θυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρακαλώ. Για την έκθεση αυτή, τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thanks Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Γενικά συμφωνούμε με τα περισσότερα σχόλια των ε, βουλευτών. Δεν επιθυμούμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Νομίζουμε ότι είναι επαρκής για τους στόχους του προγράμματος. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια γεωγραφική ισορροπία στην οποία αναφερθήκατε. Βεβαίω, συμβατότητα με τα άλλα προγράμματα είναι εκ των όνου ΚΑΝΕΦ και θα προσπαθήσουμε να την εθαρρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Τώρα, πρέπει να διευκρινίσουμε αν αφορά αυτό τις τοπικές κοινότητες και ιδιαίτερα της υπαίθρου. Εμείς θα θέλαμε να το αφήσουμε αυτό ανοιχτό. Για όλες τις τοπικές κοινότητες υπάρχουν άλλα μέσα που προσφέρονται περισσότερο ε, για πρόθεση της υπαίθρου. Εμείς θα θέλαμε να υποστηριχθούν όλες οι τοπικές κοινότητες στο συγκεκριμένο. Και αυτό ε, έχει να κάνει και με την ενδεχόμενη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. Στη δική μας πρόταση αναφέραμε κάποιες δυνατές ενδεχόμενες χρήσεις, αλλά αυτό θα το κρίνουν καλύτερα οι τοπικές κοινότητες. Ε, θεωρήσουν ότι κάπου ταιριάζει καλύτερα, είναι καλύτερη χρήση, αυτά όλα εντάσσονται στην επικουρικότητα. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς υπερβολικά ε, δεσμευτικοί και να ε, ορίζουμε με ρυθμίσεις το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Νομίζω απάντησα στις ερωτήσεις σας, δεν ξέρω αν ξέχασα καμία. Il n'y Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περάσουμε αμέσω στο τελευταίο μας θέμα που έχει να κάνει ε, πάλι με το διαδίκτυο και τη σύνδεση του ε, ε, διαδικτυακή δυσυνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Gigabit και του 5G. Η Συγητής είναι ο κύριος Ζλωτόφσκι στον οποίο και δίνω μέσο στο λόγο. Merci, la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου για τις τροπολογίες που έχουν καταθέσει. Συνεργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά με όλους τους κοιότητες ηγητές. Έχουμε έξι σχέδια συμβαστικών τροπολογιών όπου Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα από τα σχόλια των συναντέλφων. Όλες οι τροπολογίες που κάνουν λόγια για τον τουρισμό είναι θετικές, γιατί φυσικά η ανάπτυξη του τουρισμού συνδέεται άρρηκτα με τις νέες τεχνολογίες και το, δίκτυ, το ίντερνετ υψηλή ταχύτητα. Έκανα ό,τι μπορώ για να συμπεριλάβω τι τροπολογίε αυτέ, τι συμβαστικέ τροπολογίε. Πολλέ τροπολογίε ε, μιλούν για δυσανάλογα κενά και χάσματα σε ό,τι αφορά τι περιοχέ. Και για τα 5G, αλλά και για το ίντερνετ μεγάλη ταχύτητα εν γέννη. Φυσικά και πολλά πρέπει να γίνουν για να μειωθεί το χάσμα που προς το παρόν διευρύνεται Πάντως είναι ίσως καλό το ότι το παρατηρούμε ότι υπάρχει χάσμα και αν θέλουμε να το περιορίσουμε θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα, στις διαδικτυακές υποδομές και να μειώσουμε το κόστος της υποδομής. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεγόμενο blending, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή περισσότερες ε, της μιας πηγής χρηματοδότησης και να προσαρμόσουμε τα project στις πραγματικές ανάγκες. Επίσης, Συμφωνώ ότι για τη χρηματοδότηση των υποδομών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και δημόσιοι πόροι αλλά και ιδιωτικοί. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται οι συμπράξεις του δημοσιοδικού τομέα. Και ιδίω εκεί που το κέρδος είναι είτε πάρα πολύ χαμηλό είτε ανύπαρκτο. Σας παρακαλώ λοιπόν να εγκρίνετε το σημείο 4, διότι νομίζω ότι ακριβώς αυτό ε, αναφέρει ότι θα πρέπει επενδύσεις να είναι προσαρμοσμένες ε, και στους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι σημαντικό. Αν θέλουμε να φτάσουμε και στους δημόσιους επενδυτές για να επενδύσουν στις υποδομές αυτές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πείσουμε κανέναν ότι θα είναι μια υποφελή εμπορική δραστηριότητα επένδυση στα, στα δίκτυα υψηλή ταχύτητα. Μπορούμε να έχουμε αυτόνομα οχήματα, να έχουμε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τεχνολογικές υπηρεσίες, όλα εξαρτώνται από την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις εταιρείε και για τους καταναλωτές. Και η πρόσβαση αυτή θα πρέπει να δίνεται ιδίω στην ασύρματη τεχνολογία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους, ε, τους σκιώδεις συγκητές. Είχαμε πολύ ομαλή συνεργασία και παραλαμβάνω σας το να ψηφίσετε υπέρ του κειμένου αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Εσείς παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου του ΕΛΚΑ θέλω τον εισηγητή τον Κοσμά Σωτός και να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Έγινε πολύ καλή δουλειά και η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Ήδη με την εισαγωγή του ομιλία μας περιέγραψε πόσο Σημαντικό είναι αυτό το θέμα της σύνδεσης ε, και τον, του 5G ε, και για τα νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Νομίζω ανέφερε και τη μεγάλη σημασία που θα έχει ε, αυτή η νέα προσφορά για τις επιχειρήσεις, για τον τουρισμό. Θα μπορεί να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες και θα φέρει και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Μίλησε και για τη χρηματοδότηση ο εισηγητής, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για την ε, αύξηση του δυναμικού. Θέλουμε να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα διάφορα κονδύλια και πρέπει να αναπτυχθούν και νέα μοντέλα ε, για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι γιατί αναφέρθηκαν τα κενά και το χάσμα που υπάρχει, το είπε ο σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα. Υπάρχει ένα χάσμα, ιδίως για τις απομακρυσμένες ε, και ε, αγροτικές περιοχές, το είχαμε πει και στην προηγούμενη έκθεση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για αυτές τις περιοχές, να υπάρχει συνδεσιμότητα. Επίσης για το σύστημα οδήγησης, για τα αυτόνομα οχήματα, τα συστήματα ασφάλειας σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται, σε αυτά τα... στηρίζονται στη, στη σύνδεση στο διαδίκτυο γενικότερα για το σύστημα μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Η ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τις ε, ασύρματες συνδέσεις ε, πρέπει να είναι καλές αυτές οι συνδέσεις και δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια ένα τέτοια χάσματα που να επιδεινώνουν την ασφάλεια δηλαδή. Θα στηρίξουμε την έκθεση και ένα ακόμη ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία. Merci beaucoup, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Σωτόφσκι για τη γνωμοδότηση αυτή. Ήταν πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας και οι συμβιβασμοί. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες υποστηρίζουν και τις 7 τροπολογίες. Το συζήτησα με τους συναδέλφους τους, το πρότεινα και εγκρίναμε ε, αυτή την απόφαση. Συγχαρητήρια λοιπόν, και λάβαμε μάλλον αυτή την απόφαση. Το θέμα αυτό συνεχίζει την προηγούμενη συζήτηση για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται λόγος για ευφυείς μεταφορές. Είναι ένα βήμα απαραίτητο έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο ε, τα οχήματα. Γι' αυτό το σκοπό δεν αρκούν πλέον ε, οι προηγούμενες γενιές ε, ασύρματης τηλεφωνίας 3G και 4G. Αφήστε που δεν υπάρχουν πια ούτε καν σε όλη την Ευρώπη ακόμα αυτές οι συνδέσεις και μέσα σε ένα κράτος μέλος, στο ιστορικό του ίδιου κράτους για τις μεταφορές και τον τουρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Με το δίκτυο 5G θα έχουμε νέα ε, επιχειρηματικά μοντέλα και πραγματικά είναι πάρα πολλές οι δυνατότητες που ανοίγονται. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως όταν συζητούσαμε την έκθεση Τέλιτσκα, θα πρέπει να επιμείνουμε στην ψηφιοποίηση και χρειαζόμαστε 3G, 4G, 5G παντού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τέλιτσκα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψηφιακό απόγευμα, έτσι δεν είναι. Σήμερα έχουμε θεματική ε, συνεδρίαση. Καλό είναι αυτό. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζωτόφσκι. Είναι πολύ καλή η έκθεσή του και οι συμβαστικές τροπολογίες. Οι φιλελεύθεροι τις υποστηρίζουν όλες. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε δύο στοιχεία εδώ. Η πρόσβαση στην τεχνολογία 4G στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 28%, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες 75%. Φανταστείτε διαφορά. Εμείς λέμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η τεχνολογία και η επικοινωνία Gigabit. Ε, Θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε και ο ίδιος ο εισηγητής, ε, που με έχει κάπως ενοχλήσει και αισθάνομαι μια δυσφορία. Αυτό είναι η αναθεώρηση των οδηγιών και των κατευθύνων ε, γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις. Το κατανοώ αυτό, αλλά επειδή είμαι και κάπως συντηρητικός ως άνθρωπος, φοβάμαι ότι αν ανοίξουν αυτή η ασκή του αιώλου, θα οδηγηθούμε σε κάποια μη ε, κατευθυνόμενη δημιουργικότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο τομέας αυτός είναι περίπλοκος και πιστεύω ότι μπορεί να είναι υψηλό το κόστος, αλλά μπορεί να είναι και τεράστια η απόδοση. Το 2025 θα είναι πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν ισχύει αυτό, τότε είναι πραγματική ευκαιρία. Και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και τη συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου. Και από εκεί θα γίνει διαφορά. Όχι κατά ανάγκη αναθεώρηση των ισχυόντων για τις κατοικές ενισχύσεις. Βεβαίω αυτό χρειάζεται διευκρίνηση, αλλά προτιμώ το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό ήταν όμω δευτερεύον. Συμφωνώ και υποστηρίζω ε, όλες τις τροπολογίε. τροπολογίες. Ε, κυρία Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Πάντα προσπαθούμε για να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Ε, στην εποχή της πληροφορίας και η συγκεκριμένη έκθεση ε, σε αυτό αποσκοπεί. Συμφωνώ με τους συναδελφούς, δεν θα επαναλάβω τα ίδια σχόλια. Με χαρά συμπεριέλαβε κάποια δικά μας μελήματα ο εισηγητής, όπως είναι τα ευφύ συστήματα μεταφορών, αλλά η Πράσινη η Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία στηρίζουν τις συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Εύρας. Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύριος Ρεμουίνου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω χωρίς λόγο. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για την επικοδομητική τους δουλειά ως τώρα. Στην ανακοίνωση αυτή απλώς ε, αναφέρουμε τις επιθυμίες μας για το μέλλον. Η υψηλή ταχύτητα ε, διασύνδεση θα ήταν ε, σημαντική για κάθε κλάδο τη οικονομία και τη κοινωνία μα. Έχουμε θέσει κάποιου στρατηγικού στόχου στην ανακοίνωση και προσπαθούμε να δώσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα εδώ βάσει του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου που συζητιέται και στο δικό σας κοινοβούλιο και να ορίσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για το 5G. Ε, χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις εκεί όπου οι ιδιωτικές αγορές δεν μπορούν να βασιστούν απλώς ε, στα, ε, στο πόσο ε, εμπόριο και πόση ζήτηση υπάρχει. Ευχαριστούμε. Θυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, αλλά πρωτό ολοκληρώσουμε να δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή μας, στον κύριο Ζλωτοσκή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η θεωρήσει μα για το μέλλον είναι πολύ παρόμοιε, όμω αν υπάρξουν διαφορέ θα φέρουν και αύριο στην ψηφοφορία. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεγητά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κηρύξω τη λήξη τη συνεδρίαση. Όμω αύριο στι 9 ακριβώ, στι 9 με το ρολόι, θα ε, σα δω πάλι εδώ για τι ψηφοφορίε. Ε, λέω 9 και δεν εννοώ 9 και κάτι, εννοώ 9 ακριβώς και θα αρχίσουμε στην ώρα μας, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και το λέω εκ των προτέρων. Σας εύχομαι καλό βράδυ.